Έχει παρέλθει το ακαδημαϊκό τέταρτο, αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά εν μέρη η καθυστέρηση οφείλεται και στη δική μου καθυστέρηση. Αλλά ήμουν σε μία εκδήλωση. Ε, και απονομή βραβείων σε γυναίκες για επιχειρηματικότητα στην, στις αγροτικές ζώνες και τη διαβίου κατάρτιση στην Ήπεθρο. Ε, ήμουν σε αυτήν την εκδήλωση λοιπόν, γι' αυτό και καθυστέρησα λίγο. Ούτως ή άλλως όμως τις Δευτέρες πάντα ξεκινάμε με μικρή καθυστέρηση, το ακαδημαϊκό Τετάρτο δηλαδή αυτό το τέταρτο τηρούμε και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ακρόασή μας ε, με τους εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει. Πρώτος και μάλιστα ο κύριος Δεκάστρο που επίσης είναι πανεπιστημιακός μπορεί να επιβεβαιώσει ότι επιτρέπεται στα πανεπιστήμια το ακαδημαϊκό τέταρτο και άρα το έχουμε ασθενιστεί και εμείς. Καταρχήν για τα πρακτικά υπάρχουν παρατηρήσεις, φανταζόμαι ε, μάλλον για την ε, μερίστη διάταξη υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι φαντάζομαι. 20 γλώσσες διαρμηνία, μετάδοση στο διαδίκτυο τη ε, συνεδρίασή μας και έγκριση των πρακτικών τη 24 η Σεπτεμβρίου. Και τώρα περνάμε στο σεμινάριο, το εργαστήριο την, με θέμα την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020, εκτίμηση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσαμε αυτό το σεμινάριο ε, και το διαχειρίζεται ε, το τμήμα πολιτικής Β. Και η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020 έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Και έχουμε ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία αναθέτοντας ε, σε συγκεκριμένους συγκητές τις εκθέσεις επί των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το εργαστήριο θα μιλήσουμε λοιπόν για την κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2020 και θα κάνω μια εκτιμήση αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε λίγο θα σας παρουσιάσω και τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες μας σε αυτή την ακρόαση. Και μάλιστα ήδη ακούσαμε την παρουσίαση μελετών ε, και έρευνας στην Επιτροπή στις 8 Οκτωβρίου και κυρίως ασχοληθήκαμε με το θέμα της ανταγωνιστικότητας και πώς αυτή κατοχυρώνεται στην νέα κοινή πολιτική. Σήμερα θα επικεντρωθούμε κυρίως ε, στο θέμα των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και θα μιλήσουμε και για τις οργανώσεις παραγωγών, αλλά όχι μόνο. Θα διαιρέσουμε την ακρόαση σε τρία θέματα. Το πρώτο θα είναι τα στρατηγικά σχέδια μετά το 2020, ε, αξιολόγηση της ε, αρχιτεκτονικής και της διακυβέρνησης ε, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πρώτο τμήμα της ακρόαση ο εμπειρογνώμονας ομιλητής θα είναι ο κύριος Εμίλ από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας στη Σλοβενία. Το δεύτερο τμήμα της ακρόασης, το δεύτερο θέμα θα είναι η στήριξη της ΚΑΠ μετά το 2020 η αξιολόγηση της μελλοντική δομή των άμεσων ενισχύσεων και των παρεμβάσεων στην αγροτική ανάπτυξη υπό το φως των προκλήσεων ε, στη γεωργία και το περιβάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα ακούσουμε τον δόκτωρα Ρολ Γιόγκενιλ από το, από Πανεπιστήμιο του Βάγγενιγκεν στις κάτω χώρες. Καλώς ήρθατε και εσείς κύριε Γιόγκενιλ. Και το τρίτο τμήμα της ε, δημόσιας ακρόασης ε, θα ασχοληθεί με την ΚΑΠ μετά το 2020 και τις λύσεις για να βελτιωθεί, να βελτιωθεί η αλυσίδα αξιών στα τρόφιμα. Εδώ ε, θα μας κάνει την ομιλία ο Δόκτωρ Τόμας Γκαρσία Ασκάρατε από το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ισπανίας. Θα δώσω το λόγο για ένα τέταρτο στον κάθε μας καλεσμένο και μετά τις ομιλίες των εμπειρογνωμόνων θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές μας, την κυρία Εράν, την κυρία Μίλλερ και τον κύριο Αντριέ. Μετά αυτή, αυτό το πρώτο γύρο με παρατηρήσεις και ερωτήσεις των εισηγητών θα ξαναδώσω το λόγο για άλλο ένα τέταρτο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν και αν το επιτρέπει ο χρόνος θα οργανώσουμε και δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων. Κυρία Κιλέρα μου ζήτησε το λόγο. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι η διεθνή ημέρα της γυναίκας στην Ήπεθρο και εμείς είμαστε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν μπορεί η Επιτροπή μας να μιλάει υπόψη την ιδιαίτερη ανάλυση που χρειάζεται η θέση της γυναίκας στην Ήπεθρο ε, για τη γεωργία και για τις αγροτικές ζώνες γενικώ. Οπότε θα ήθελα αυτό να αναφέρω κατά την έναρξη της συνεδρίασής μας σήμερα γιατί και προσωπικά αλλά και η πολιτική μου ομάδα θα ήμασταν υπέρ μιας κοινή γεωρικής πολιτικής με μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών. Να φαίνεται περισσότερο το πρόσωπο της γυναίκας ή να είναι πιο εμφανής ο ρόλος των γυναικών στις αγροτικές ζώνες και στην ύπεθρο γενικώ. Γι' αυτό και ζήτησα το λόγο κατά την έναρξη της συνεδρίασης για να τονίσω ότι σε μια τόσο σημαντική μέρα και με τόσο σημαντική εκδήλωση δεν, δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα να περάσει απαρατήρητο. Κυρία Αγγιλέρα, σας είμαστε ευγνώμονες που το επισημάνατε. Εγώ στην αρχή που σας είπα ότι ήμουν σε μια εκδήλωση με απονομή βραβείων από την Κόπα Κοζέκα, ε, το θέμα ήταν ακριβώς οι γυναίκες στην Ήπεθρο αλλά και εσείς ε, εντάξετε το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο αυτό που είπατε και ο ρόλος των γυναικών και η παρουσία των γυναικών στην ύπεθρο και στις αγροτικές ε, ζώνες χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Και χαίρομαι που έχουμε πολλές γυναίκες στην αίθουσα γιατί Βλέπω ότι και στην Επιτροπή μας έχουμε πολλές γυναίκες που ασχολούνται με τα θέματα της γεωργίας, τα αγροτικά ζητήματα. Έτσι, έστω και έμεσα έχουμε παρουσία γυναικών στα θέματα αυτά. Πέραν της πραγματικής παρουσίας των γυναικών στη γεωργία και στην Ήπεθρο. Σας ευχαριστούμε κυρία Αγγιλέρα για την επισήμανση. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σεμινάριό μας, στο εργαστήριό μας. Δίνοντα το λόγο για ένα τέταρτο στον κάθε εμπειρογνώμονα. Ευχαριστώ. Μια στιγμή. Και ο κύριος Φλάναγκα ζήτησε το λόγο. Ναι. Ε, θα προτιμούσα να μην είμαι υποχρεωμένο να πάρω το λόγο. Ε, ήθελα πολύ να έρθω να ακούσω αυτό το εργαστήρι και σηκώθηκα με χαρά το πρωί. Αλλά προς πρέπει να ε, σημειώσω την απογοήτευσή μου όσο και την αηδία μου για την ισχνή παρουσία των συναδέλφων. Την τελευταία φορά είπαν οι συναδέλφοι ότι ήταν δύο πολύ ε, ε, φορτωμένες μέρες. Εγώ μίλησα με τον πατέρα μου και μου είπε «Ξέρεις τι Ελληνίδη πώς δίνει αυτό». Δηλαδή μετά τη δεύτερη μέρα έχουν κουραστεί. Σήμερα είναι πρώτη μέρα. Δεν φταίει κανένας παρόν αλλά είναι ύβρι προς του ανθρώπου που έρχονται και προ τα παιδιά μου που δεν τα βλέπω γιατί έρχομαι στη δουλειά μου όταν οι συνάδελφοι ε, απαξιούν να πατήσουν στη συνεδρίες. Σα ευχαριστούμε κύριε Φλάναγκαν. Ε, όντως δίκαιη η παρατήρησή σας. Και τις Δευτέρες έχουμε συχνά πρόβλημα με την προσέλευση αλλά οι πληροφορίες που θα ακούσουμε από τους εμπειρογνώμονες μας θα φτάσουν μέσω των βοηθών των συνεργατών και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Πάντως, όντως, εύστοχη παρατήρηση και περνάμε στο εργαστήριο και δίνω το λόγο στον πρώτο μας εμπειρογνώμονα, τον κύριο Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, συνάδελφοι, κληθήκαμε να αξιολογήσουμε το σχεδιασμό της, του νέου στρατηγικού σχεδίου της κοινή γεωργικής πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στον τίτλο 5. Το Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα τελεχώνεται από διεθνείς οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες. Ε, η ανάλυση βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση του νέου προτύπου απόδοση ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής, τον υπολογισμό των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο. Επιτρέψατε μου να σας παρουσιάσω τα κύρια πορίσματα αυτής της μελέτης και ιδιαίτερα στις συστάσεις πολιτικής. Η μελέτη βασίζεται στην χρήση διαφόρων συμπληρωματικών μεταξύ τους πηγών. Πρώτον, ε, συστηματική ε, έρευνα των πληροφοριών αυτών. Έχουμε μελέτες από ομάδες ε, πίεσης και για τα κράτη-μέλη είναι προφανές ότι δεν είναι θέμα έρευνας, αλλά και άρα είναι δύσκολο να προβούμε σε αντικειμενικές αναλύσεις, οπότε αναπτύξαμε ένα επόμενο βήμα, ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο είχαμε πολύ, καλές, ε, πολύ καλή ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους και από τους γεωργούς και από την ε, τομέα της διοίκησης και από τους ερευνητές. Τρίτον, βασιζόμαστε στο πλαίσιο λήψης πολιτικών αποφάσεων και χάραξη πολιτικής. Γιατί, γιατί αυτό το πλάνο πλαίσιο πολιτικής θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές επιστημονικές ε, αποδείξεις και στοιχεία. Στην πράξη, ωστόσο, παρακολουθούμε εκείνους τους ε, ε, επιστήμονες που αναφέρουν ότι η χειραγώγηση, τα λόμπι, όλα αυτά είναι ένα σύστημα τέτοιο που είναι πολύ δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή. Είναι περιορισμένη λοιπόν η προσέγγιση και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη όταν ε, αξιολογούμε τις προτάσεις. Εν γέννη, το νέο πρότυπο για την αποδοτικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σωστό βήμα ε, προς την κατεύθυνση της διακυβέρνησης ε, από τον δημόσιο, δημόσιο τομέα και ωστόσο η το προτινόμενο μοντέλο βασίζεται στο καθιερωμένο πρότυπο της ανάπτυξης υπαίθρου και βασικά καλύπτεται από το ίδιο σύστημα διακυβέρνησης. Οπότε περιλαμβάνει διάφορα από τα προβλήματα του ισχύου του συστήματος. Οι κίνδυνοι συνδέονται με τις πιο αδύναμες δομές, το διοικητικό φόρτο, τον ελπίσει σχεδιασμό από πλευρά των κρατών μελών και ο κίνδυνο είναι να μειωθούν τα στάνταρ ή να υπάρξει μια προσπάθεια προς την μείωση των στάνταρ. Η μελέτη μας ε, λέει ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις θα οδηγεί, που στόχο έχουν να οδηγήσουν σε μια πολιτική με βάση τα αποτελέσματα. Ωστόσο, εμείς βλέπουμε πως τα κράτη-μέλη ε, είναι απρόθυμα να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες και τονίζουμε τη συστημική αδυναμία στη λογική παρέμβαση μέσα στο πλαίσιο του νέου μοντέλου. Κάποια παραδείγματα. Τρεις στόχοι για το περιβάλλον και οι σχετικοί δείκτες δεν συνδέονται άμεσα με ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι προτάσεις αυτές επίσης δεν είναι σαφείς όσον αφορά το, την μέθοδο ποσοστοποίησης της βασικής ε, ε, γραμμής. Τα, ε, δε, η δε τεχμηρίωση και οι αναλύσεις για έγκριση από την Ένωση είναι ελλειπή. Το σημερινό σύστημα και τα, μέτρα σχεδιασμού είναι περιοριστικά. Τα κράτη-μέλη μπορούν μόνο να επιλέξουν κάποια μέτρα και να τα υιοθετήσουν. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού αφήνεται, ε, επαφείται στις ικανότητες των κρατών μελών, στις δυνατότητες των κρατών μελών. Ο μονός στόχος είναι να μπορεί να μετρηθεί η απόδοση. Οι εθνικές προτεραιότητες δεν ε, προκύπτουν από κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητος τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η διαδικασία που συνδέεται με την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου είναι ο μόνος μηχανισμός που μπορεί να εξασφαλίσει ένα ε, φιλόδοξο στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ποιοτική αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων που θα πρέπει να περιλαμβάνουν ικανοποιητικό και ισορροπημένο επίπεδο ε, διαβούλευση ανάμεσα στου ενδιαφερόμενου φορεί και τι άλλε δημόσιε αρχέ. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα προσχέδια σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίση, θα πρέπει να είναι πιο τυποποιημένη η διαδικασία ε, και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψει των ε, ενδιαφερομένων φορέων και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ε, ε, νομιμοποιείται το έγγραφο αυτό. Ο κίνδυνος προκύπτει βασικά από την ίδια στις δυνατότητες των διαφόρων φορέων στα κράτη-μέλη. Δεδομένου ότι ε, μέχρι στιγμής ε, οι προσεγγίσει ήταν ανά μέτρο. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν αρκετή εμπειρία στο να προγραμματίζουν διάφορα μέσα της κοινή γεωργική πολιτικής με ολοκληρωμένο τρόπο και γι' αυτό προβλήματα στην επικουρικότητα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικό διοικητικό φόρτο στα κράτη-μέλη. Οπότε η ανάπτυξη ε, δυνατοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογή ε, θα είναι πρόκληση για πολλά κράτη-μέλη και ιδιαίτερα για εκείνα τα, τα κράτη-μέλη που είναι μικρότερα και για τα κράτη-μέλη που θα μπουν στην Ένωση μετά το 2024. Γι' αυτό και χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και προετοιμασία, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρχουν διαφορέ σημαντικέ στην εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Πράγμα που θα σημάνει ε, πρότυπα στα κράτη-μέλη και αποδυνάμωση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλιστικές δικλίδες, ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών που θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση της προόδου του ε, σχεδίου του εκάστοτε σχεδίου. Θα πρέπει αυτά όλα να είναι μέρος της διαδικασίας έγκρισης. Κάτι ακόμα, η, ε, ένας προϋπολογισμός ε, προενταξιακός θα μπορούσε να διευρύνει τη ε, στοιχεία προϋπολογισμός που θα μπορούσε να ε, ισχύσει και για τον πρώτο πυλώνα τη κοινή γεωργική πολιτική. Η παρακολούθηση και η διαδικασία αξιολόγηση θα πρέπει να οριστούν πιο συγκεκριμένα και να βελτιωθεί η ποιότητά τους σε όλα τα τμήματα του κύκλου ε, πολιτικής. Η επόμενη περίοδος θα είναι περίοδος εκμάθησης όπου θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η ποιότητα των πηγών των στοιχείων στα κράτη-μέλη και στα ευρωπαϊκά όργανα δηλαδή GRC, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Περιβάλλον, Eurostat, όλοι αυτοί ε, θα έχουν ρόλο να παίξουν εδώ. Τονίζουμε λοιπόν το ρόλο των στοιχείων, των δικτών, των, των γνώσεων και των αναλύσεων για πιο αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν ε, ε, στοιχειοθετημένες ε, πηγές ε, δεδομένων. Μία από τις ιδέες είναι να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα με ανοιχτή πρόσβαση για όλα τα στρατηγικά σχέδια και αναλύσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Γεωργία κάθε φορά. Κάνουμε και κάποιες προτάσεις λοιπόν για τροποποίηση του προτινόμενου κανονισμού. Καταρχάς να ισχύει η αρχή της μη οπισθοδρόμησης, δηλαδή να έχουμε ένα σχετικά ε, δίκαιο μερίδιο στήριξης για τις κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Δεύτερον, να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι ποσοτικοί στόχοι με βάση την νομοθεσία και τις δεσμεύσεις και επίσης ε, δίνουμε κάποιες ιδέες σε σχέση με τη νομοθετική πρόταση η οποία χρειάζεται να διακάνει σαφέστερη διάκριση ανάμεσα στους κοινού και τους εθνικούς στόχους γιατί εδώ βασικό θέμα είναι οι στόχοι που σχετίζονται με τα έσοδα και την κοινωνική κατάσταση στις περιοχές της υπαίθρου. Δεύτερον, να ενισχυθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς στη διάρκεια της διαδικασίας κοινή λήψη αποφάσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν μέσα, μάλλον να αποσαφινιστούν περισσότερο. Στο 206, άρθρο 206, προτείνουμε να προσθεθεί κάτι για την φιλοδοξία και την δυνατότητα υλοποίησης των εθνικών στόχων ε, για την βελτίωση των στοιχείων, επί τη βάση των υπερχόντων όμως δεδομένων. Δεύτερον, ένας ε, κατάλογος προτάσεων ε, περιλαμβάνει και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του συστήματος συντονισμού με τα περιεχόμενα του τρίτου παρατήματος, ε, τις εταιρικέ σχέσεις δηλαδή και την καθολική προσέγγιση. Και επόμενη παρατήρηση αφορά την απλοποίηση που πάνω κάτω απευθύνεται στα κράτη-μέλη, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και η συσχέτιση με τους στόχους της Ένωσης και να συμπεριληφθεί υποχρέωση για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και η συμπερίληψη ε, Έκθεση αντικτύπου στη, μέσα στο σύστημα παρακολούθησης γιατί πιστεύουμε πως μόνο οι δείκτες αποτελεσμάτων που, έχουν, που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις δεν αρκούν για να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα την κατάσταση και να έχουμε ένα φιλόδοξο ε, σχέδιο. Έπειτα, το υποχρεωτικό κομμάτι της ε, έκθεσης θα πρέπει να βελτιωθεί και ποιοτικά και ποσοτικά και προτείνουμε αυτό να γίνει και από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, θα πρέπει να Ε, θεσπίζονται βάσεις δεδομένων και αναλυτική ε, στήριξη για τα, ε, για τα προγράμματα κάθε φορά. Για την περίοδο λοιπόν 2021 μέχρι 2027 θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη περίοδο ανάπτυξης για το στρατηγικό σχεδιασμό της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά όχι μεγάλη αλλαγή των μέτρων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ιδιαίτερα βελτιωμένα στοιχεία, γιατί οι αλλαγέ είναι τόσο βαθιές που θα πρέπει να γίνει μια πιο μακροπρόθεσμη ανάλυση και έκθεση με, βάση τη, δημιουργία συστημάτων οι συνομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουν τι περιμένουν από την πολιτική άποψη από αυτό το νέο μοντέλο απόδοσης. Εάν στόχο είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και πολιτική ευθύνη, θα πρέπει αναλόγως και να ενεργήσουν ώστε να διευκολύνουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, ε, προσέγγιση με βάση τις, ε, τα στοιχεία, τα δεδομένα και ε, ανταγωνισμό ανάμεσα στις χώρες. Το στρατηγικό λοιπόν αυτό σχέδιο θα πρέπει να είναι ένα βήμα προς την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των πολιτικών αυτών μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, εμείς ευχαριστούμε κύριε Ριάβετς. Περνάμε τώρα στον κύριο Γιον Γκενίλ από το Οικονομικό Συμβούλιο Έρευνας του Πανεπιστημίου Βαγγένιγκεν. Για ένα τέταρτο κι εσείς. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, να μιλήσω ε, για τις προτάσεις ε, σχετικά με το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα επικεντρωθώ στην ανάπτυξη πέθρου στις άμεσες πληρωμές και στα αντίστοιχα θέματα που είναι ο τίτλος 3 των νομοθετικών προτάσεων. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά το εισόδημα των γεωργών, το περιβάλλον και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όλες αυτές οι προκλήσεις και τα προβλήματα διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια. Είναι πολύ μεγάλη ετερογένεια, όπως λέμε. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Χρειαζόμαστε κάποια μέτρα ανάλογα με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχει η κάθε περιφέρεια για να δούμε πώς ε, μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ανταπεξέλθουμε. Ευθύς εξ αρχής έχουμε διαπιστώσει ότι χρειάζεται πολύ στοχευμένη παρέμβαση και πολιτικές κομμένες και ραμμένες ε, στα μέτρα της εκάστοτε πραγματικότητας. Θέλω να το πω από την αρχή αυτή. Η επικουρικότητα πρέπει να κυριαρχήσει και θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ακριβώς για να σχεδιάσουμε καλύτερα τις πολιτικές. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε στην ε, ε, αρχή της επικουρικότητας. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στο τίτλο 3 για να δούμε ποια είναι τα μέσα που προβλέπονται για τις παρεμβάσεις ε, σε σχέση με τη σημερινή κοινή γεωργική πολιτική. Δηλαδή θα δούμε πώς λειτουργούν σήμερα τα πράγματα, αν θα χρειαστούν νέα, αν είναι αντίστοιχα, τι μπορούμε να δούμε από τη βιβλιογραφία, τι μπορούμε να δούμε από το δυναμικό που έχουν και από άλλες εμπειρίες ε, στην πράξη, στη θεωρία. Αν, υπάρχουν αν υπάρχουν μάλλον πληροφορίες που μας βοηθούν για να επιλέξουμε κάποιο μοντέλο, για να εφαρμόσουμε κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις, για να κάνουμε και προτάσεις όσο και συστάσεις. Θέλω να τοποθετήσω λίγο τη συνεισφορά μου για να καταλάβουμε το πλαίσιο. Βλέπετε εδώ μια γραφική παράσταση. Βλέπετε τον κάθετο άξονα, το ύψιλο ας πούμε, που είναι το εισόδημα των ε, γεωργών. Ε, ο άξονας οριζόντιος στο Χ είναι το περιβάλλον και η βιοπικιλότητα. Και έχουμε και ένα διαγώνιο ε, άξονα ε, αυτό που είπε ε, προηγουμένως ο συνάδελφος αφορά τις εξελίξεις. Ε, κοιτάξτε δηλαδή το πράσινο τόξο από το status quo που είναι η σημερινή κατάσταση προς το επιθυμητό σημείο. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στα τόξα που βλέπετε εδώ, τα διάφορα μέσα και εργαλεία που υπάρχουν για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στους διάφορους στόχους μας. Αυτό είναι το πλαίσιο που ονομάζεται Free είναι, ένας, ε, ε, είναι οικονομολόγοι αυτοί που έχουν βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ από το, ε, τις κατοχώρες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πλαίσιο ε, όταν υπάρχουν ειδικοί και πολλαπλοί στόχοι που θα πρέπει να είναι ορισμένο και το ανέφερε και ο προηγούμενος συνάδελφος. Ας περάσουμε λοιπόν στις άμεσες πληρωμές, ενισχύσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα μέτρα για την ανάπτυξη πέθρου και τέλος θα κάνω κάποιε προτάσει και συστάσεις για βελτίωση και συζήτηση. Πρώτον, για τις άμεσες πληρωμέ. Η ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματο υποφέρει από μεγάλες ανισότητες. Γνωρίζουμε ότι το 81% των αμέσων ενισχύσεων πηγαίνουν στο 20% των αγροτών σήμερα και αυτό ε, μπορείτε να μου πείτε ότι ισχύει γιατί δεν είναι παντού ε, εξισωμένες οι άμεσες πληρωμές. Αν είχε γίνει αυτή η εξίσωση, τότε θα λέγαμε ότι 86% των ενισχύσεων θα πήγαιναν στο 20% των γεωργών. Άρα αυτό το επιχείρημα εντείνει το θέμα της ανισότητας. Άρα χρειαζόμαστε καλύτερα κριτήρια που να είναι πιο πολύ προσανατολισμένα στις ανάγκες ε, της εκάστοτε ε, κατάστασης για να είναι πιο στοχευμένες οι άμεσες πληρωμές και να έχουν μια πιο συγκεκριμένη ε, παρέμβαση και στόχο. Η νέα λοιπόν κοινή γεωργική πολιτική ε, βασίζεται στα εκτάρια, στα, στα στρέμματα ε, και όχι στις ανάγκες των γεωργών. Άρα δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα 100%. Τα λύνει σε κάποιο βαθμό γιατί υπάρχει και κάποια ενίσχυση περιορισμένη με ανώτατο όριο και το ελεκτικό συνέδριο πρόσφατα σε μια έκθεση έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά, ένα νέο στοιχείο ε, είναι τα οίκο ε, σχήματα που προτείνονται. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον μέτρο που επιτρέπει και διευρύνει ε, τις δράσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του κλίματος. Δηλαδή, η φιλοσοφία είναι ότι το δημόσιο χρήμα εξυπηρετεί ε, το δημόσιο συμφέρον και είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά είναι ακόμα πολύ ε, ασαφές το πώς τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν όλα αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Ε, αυτή τη στιγμή δεν ορίζεται πολύ σαφώς από την νομοθεσία πώς θα εφαρμόστη εμείς λέμε ότι υπάρχει χώρος διεύρυνσης και του πεδιοφαρμογής ε, και της κάλυψης των ε, σχημάτων αυτών. Τώρα είναι στρεματική ενίσχυση για τις ε, προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες. Αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί αυτό και να συνδεθεί και με κάποιες δράσεις. Στη νέα βασική ε, γραμμή, ας πούμε, έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης ε, των γεωργικών εφοδίων. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο για τους αγρότες, αλλά στο οικολογικό σχήμα να αξιολογείται και να λες στον αγρότη ότι εάν με αυτό το μέσο προσπαθείς να βελτιώσεις την κατάστασή σου, το περιβάλλον και το κλίμα, τότε θα έχεις και κάποια μια ανταμοιβή με βάση ένα point system. Άρα ε, θα ε, εξαρτηθούν οι ενισχύσεις από την απόδειξη. Βέβαια χρειάζεται μια ευελιξία ε, στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Άλλο παράδειγμα. Αυτό το εργαλείο διαχείριση των εφοδίων είναι χρήσιμο για τους αγρότες, αλλά πρέπει να μάθουν να το χειρίζονται. Άρα, αν κάποιος αγρότης σε ένα σεμινάριο, μια κατάρτιση για τη συγκεκριμένη αυτή δράση, θα πρέπει να, να αμείβεται επίσης. Άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις άμεσες ενισχύσεις είναι η οροφή που ε, έχει ε, προταθεί το κάπινγκ. Κατά την άποψή μας αυτό δεν θα έχει σχεδόν καθόλου ε, αποτέλεσμα στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα. Δηλαδή από τις άμεσες πληρωμές ο αγρότης θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεί όλο το, όλα τα έξοδα ε, προς το προσωπικό της εκμετάλλευσης αλλά να αφαιρεί και το νοητό εισόδημα τους μισθούς της οικογένειας που δεν αμείβεται από αυτή τη γεωργική δραστηριότητα. Οπότε τότε δεν θα υπήρχε κανένα κάπινγκ ή θα ήταν πολύ περιορισμένο. Άρα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό το μέτρο. Επίσης, η ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση εισοδήματος ε, για τη βιωσιμότητα ε, έχει αναφερθεί και στη σημερινή κοινή γεωργική ε, πολιτική. Δηλαδή είναι πληρωμές που βοηθούν ειδικού τομείς που είναι σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, ας πούμε, σε κάποιες περιφέρειες που είναι σε ύφεση ή σε παρακμή. Και πάλι θα πρέπει να είναι στοχευμένη η εφαρμογή και εμείς τι προτείνουμε όχι πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τη σημερινή κοινή γεωργική πολιτική, αλλά από την εμπειρία του συστήματος έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή η υποστήριξη, έτσι όπως δίνεται η ενίσχυση εισοδήματο, δεν είναι αρκετά διακριτική, δηλαδή γίνεται αδιάκριτα με γενικό τρόπο. Για ποιο λόγο ε, ο οι Γάλλοι γαλακτοπαραγωγοί στο σύνολό τους χρειάζονται άμεσε ενισχύσει. Μπορεί αυτό να ισχύει για κάποιες περιφέρειες, για κάποιες ορεινέ περιοχές, αλλά όχι γενικά όλος ο γαλακτοκομικός τομέας στη Γαλλία. Πάρτε ενίσχυση. Υπάρχει και αρχή της εξειδίκευσης της παραγωγής. Και στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θέλουμε και μια αποτελεσματική παραγωγή, δηλαδή τουλάχιστον να λαμβάνει υπόψη το κόστος. Βέβαια, σε κάποιες περιφέρειες, επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος, δεν συμφέρει η παραγωγή. Ενώ σε άλλες περιφέρειες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μια ισορροπία. Στοχευμένη στήριξη του εισοδήματο μένα, αλλά και ε, στήριξη της αγοράς. Μετά, έχουμε και κάποιες ανησυχίες ως προς την ανταγωνιστικότητα και τους ε, ίσους όρους παιχνιδιού και ανταγωνισμού. Αυτό μιλάμε για ενισχυμένη ερεσιμότητα, δηλαδή και με κάποια ευελιξία δεν λέω, ενισχυμένη ερεσιμότητα ε, ορίζει ποια είναι η βασική γραμμή που θα ισχύει για όλους και πέρα από τη ε, διασταυρωμένη συμμόρφωση που ισχύει και σήμερα στην ΚΑΠ υπάρχουν κάποια στοιχεία του πρασινίσματος ας πούμε που συμπεριλαμβάνονται αλλά υπάρχει κάποια διακριτική ευκαιρία για τα κράτη-μέλη, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν ποια θα είναι αυτή η βασική γραμμή, που μπορεί να είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Αυτό έχει να κάνει με το θεμητό ανταγωνισμό και τους ίσους όρους. Σε πάση περιπτώσει, το γράφουμε, δεν είναι τόσο σημαντικό. Μετά, ε, έχουμε τις πληρωμές για τα οίκο ε, σχήματα. Είναι στρεματική ενίσχυση αυτή και μπορεί να καλύψει ένα κόστος εισόδημα από λεσθέν ε, μπορεί να είναι επιπλέον της τρεματικής ενίσχυσης. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Δίνουμε μια επιπλέον αμοιβή στους ε, γεωργούς που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Για το κλίμα τώρα υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και από τα λεγόμενα οίκο-σχήματα είναι αρκετά περιορισμένη η πρόταση στην καθοδήγηση που δίνει στα κράτη-μέλη για το πώς θα το εφαρμόσουν αυτό. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό κάτι δεν το περίμενα καθόλου από την πρόταση. Τώρα για την πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου. Οι αλλαγέ είναι σχετικά περιορισμένες, το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Έχουμε ένα νέο μοντέλο απόδοσης ε, αγροπεριβάλλον, κλίμα και άλλες ε, δεσμεύσεις διαχείρισης ισχύουν και σήμερα στην ΚΑΠ. Και αυτό καλύπτει ε, ένα ευρύ φάσμα στόχων. Εννέα συγκεκριμένους στόχους της ΚΑΠ και αν τους παρατηρήσετε και τους μελετήσετε θα δείτε ότι όλα αυτά τα μέσα και εργαλεία μπορούν να διορθώσουν το στόχο. Δηλαδή και τα οικοσχήματα και αυτά τα μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα είναι παρεμφερή. Και πάνω κάτω επαρκούν για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν παντού ε, τους στόχους κοινή γεωργικής πολιτικής. Γενικά υπάρχει ένας γενικός κανόνας που λέει ότι για να φτάσεις σε ένα στόχο πρέπει να έχεις αρκετά μέτρα προς το στόχο αυτό. Αυτό ισχύει. Άλλο σημαντικό. Η υποστήριξη των επενδύσεων. Έτσι αλλάζει και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας. Ενώ στις άμεσες πληρωμές αν δείτε την εξάρτηση των αγροτών από αυτές είναι πάνω από 40%. Ε, δεν θέλουμε οι στοδίνικες να εξαρτώνται από τις ενισχύσεις οι αγρότες. Θέλουμε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να αυτό εξυπηρετούνται οικονομικά. Ε, αυτό σημαίνει μακροχρόνια βιωσιμότητα. Τώρα, οι ρυθμίσεις για τους νέους αγρότες ε, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ και με τις ανάγκες. Εντάξει, το ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους νέους αγρότες, αλλά σε κάποιες περιφέρειες είναι κατακαιρματισμένη η δομή η ίδια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είναι πάρα πολύ μικρές οι εκμεταλλεύσεις. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ανανέωση, η μεταβίβαση ε, της εκμετάλλευσης σε ένα νέο αγρότη, αλλά η ανεδιάρθρωσή της. Επίσης υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορούμε να συνδυάζουμε με διάφορες μορφές ε, αλληλασφάλισης και τα λοιπά. Επίσης συνεργασία και γνώση και τεχνογνωσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την καινοτομία να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν τις γνώσεις και ε, να συνεργάζονται οι αγρότες. This, let Τούτων λεχθέντων έρχομαι και συνοψίζω στις ε, συστάσεις. Πρώτον, ως προς τις οροφές, το ανάτατο όριο αυτό το κάπινγκ, υπάρχει μια φόρμουλα που κάνει τον υπολογισμό 50.000 ε, ευρώ το σύνολο, το, το όριο των πληρωμών. Μετά όμως αφαιρούνται οι μισθοί. Εγώ προτείνω να υπάρχει ένας ε, συστηματικός τρόπος υπολογισμού ε, του πόσο είναι το εργατικό κόστος ε, σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Ας πούμε 50 στάνταρ μονάδες αναεργαζόμενο. Άρα, ας πούμε, η μέση εκμετάλλευση χρειάζεται δύο γεωργικούς εργάτες και τα κριτήρια να βασίζονται σε αυτό και όχι στον πραγματικό αριθμό εργαζομένων σε μια γεωργική εκμετάλλευση που μπορεί να είναι μεγάλος. Ιδιαίτερα αν παραμείνει το εργαλείο του κάπινγκ έτσι το νότο του ορίου όπως προβλέπεται σήμερα μετά την αφαίρεση των μισθών συμφέρει το γεωργό να προσλάβει πολύ προσωπικό στην ε, εκμετάλλευση. Εγώ προτείνω λοιπόν να γίνει ένα μονάδα εργασίας και εργαζομένου. Και αν αυτό το μέτρο του κάπινγκ χρησιμοποιείται για να εξισώνεται ε, το εισόδημα, τότε θα παίρνουν λεφτά οι αγρότες για άλλους λόγους, ας πούμε για οικολογικά, για το κλίμα, για το περιβάλλον. και δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο γιατί δεν είναι εισοδηματική ενίσχυση του αγρότη και των εργαζομένων του αλλά πηγαίνει σε άλλους σκοπούς περιβαλλοντικούς και λοιπούς. Άρα εγώ προτείνω ε, να είναι προαιρετική αυτή η σύνδεση με την ε, έκπτωση των μισθών και να προσθεθούν και άλλοι στόχοι να μην είναι μόνο η ενίσχυση του εισοδήματος. Τώρα, περιορισμός επίσης της παραγωγής. Ας πούμε το 1 τρίτο της παραγωγής να ε, ε, δέχεται άμεσα ενισχύσεις. Αν ένας ολόκληρος κλάδος ε, σε μία χώρα ζητάει συνδεδεμένη ενίσχυση, τότε αυτό είναι κατάχρηση του μέτρου. Σε ό,τι αφορά τώρα για τους νέους αγρότες, είναι καλή η πρόταση, αλλά θα πρέπει να ε, ικανοποιείται το κριτήριο της βιωσιμότητας πολύ περισσότερο. Και υπάρχει και λόγος. Έχουμε το θέμα της συμβατότητας με τον ΠΟΕ Και τώρα έρχομαι στα οίκο σχήματα, οίκο schemes. Στη σημερινή ΚΑΠ το 30% των άμεσων πληρωμών πηγαίνουν στο πρασίνισμα, το greening. Αυτό είναι πολύ ασαφές, πολύ γενικό και αόριστο και δεν συνδέεται με συγκεκριμένες προσπάθειες που καταβάλουν οι αγρότες. Τώρα αλλάζει το σύστημα αυτό και δεν έχει και ασφαλιστική δικλίδα. Θα πρότεινα να μπει μια ασφαλιστική δικλίδα, ένα ποσό, όχι 30% αλλά 50%. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν θα είναι απλώς υποχρεωμένα να το εφαρμόζουν, αλλά θα πρέπει να το συγχρηματοδοτούν κατά το ίμιση. Και μετά, αντί να είναι στρεματικές ενισχύσεις συνδεόμενες με την επιφάνεια, να συνδέονται με κάποιες δράσεις. Ε, κατάρτιση, α πούμε, ή κάποιοι αγρότες που εθελοντικά συμμετέχουν σε κάποια συστήματα πιστοποίησης και ιδιωτικά σήματα για την ευζοία των εκτρεφόμενων ζώων κτλ. Όχι πράγματα που να τους επιβάλλει η αγορά, αλλά εθελοντικά να προχωρούν σε κάποιες κινήσεις που θα είναι καλές για την κοινωνία, μπορεί να επιβραβεύονται με αυτό το point system και με περισσότερες ενισχύσεις. Για την ανάπτυξη, την αγροτική, είναι πολύ σημαντικές οι ε, επενδύσεις. Αν δείτε όμως τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο ως προς τη διαφάνεια και την επιλογή των έργων, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σοβαρές ε, δυσλειτουργίες όσο και ανομαλίες και χρειάζεται βελτίωση, ίσως και μεγαλύτερη καθοδήγηση από την νομοθεσία. Υπάρχουν και κάποιες επενδύσεις μη παραγωγικές όπως είναι η ανανέωση ε, των στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης, η καινοτομία πάρα πολύ σημαντική και η υποστήριξή της. Αν κοιτάξετε τις εταιρείες εκτός γεωργίας ας πούμε, ο προϋπολογισμός τους για την έρευνα είναι περίπου στο 5% και πολλοί καινοτόμες έχουν πολύ πιο ψηλά. Ε, σε κάποιες μελέτες που διάβασα για την ανάλυση αυτή είδα ότι στη Γεωργία είναι το 1% μόνο που πηγαίνει στην καινοτομία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κατόφλι και πάλι ως ασφαλιστική κλίδα ότι κοιτάξτε κύριε ο προπολογισμό σας για την καινοτομία θα είναι τόσος τουλάχιστον. Uh, λοιπόν, τα είπα για τον ΠΟΕ που γενικά ισχύει αυτό για διάφορα κεφάλαια και χρειάζεται ε, διευκρίνηση, διαχείριση του κινδύνου επίσης καλύτερη, χρειάζεται να δοθεί προσοχή. Προβλέπετε μεν, εντάξει. Για τη διαχείριση του κινδύνου επίσης, στις, στα σημερινά μέτρα βλέπουμε ότι είναι κάτω των αναγκών και κάτω των προσδοκιών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν μήπως θέλουν να επιβάλλουν ως υποχρεωτική κάποια ασφάλιση. Γιατί αν δεν είναι ασφαλισμένοι οι αγρότες, θα κληθούν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια, να καλύψουν ε, το ρίσκο όταν υπάρχει ένας κίνδυνος. Άρα μήπως να τους υποχρεώνουν να κάνουν και ασφάλειες. Then finally on level playing field. Για ε, τους ίσους κανόνες παιχνιδιού τώρα και τον ανταγωνισμό. Το είπα και προηγουμένως. Ε, ε, και για τα διάφορα οικολογικά σχήματα και για τις άμεσες πληρωμές και παντού, το είπα προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχουν οι ε, ίσοι συγκανόνες. Τέλος. αξιολογήσεις. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αποτελεσματικός μάλλον. Ε, ε, φαίνεται αυτό από τις αξιολογήσεις. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος. Το μερίδιο ε, των χρημάτων που πηγαίνουν στο δεύτερο πυλώνα κινδυνεύουν να μετατεθούν και πάλι στον πρώτο και θέλουμε αυτό να το αποφύγουμε. Τελευταίο και κλείνω. θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση ότι η βιοπικιλότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο της βιώσιμης γεωργίας. Αυτά και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστούμε. Και... Παρακαλώ τον τρίτο μας καλεσμένο, τον εμπειρογνώμων ε, καθηγητή Τόμας Γκαρσία Καράτ να τηρήσει το χρόνο που δικαιούται, το τέταρτο δηλαδή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Mm. Mm. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά. Ε, για να δουλέψουν και οι υπόλοιπε καμπίνες γιατί παρά είναι εύκολα τα πράγματα για την Ιταλική καμπίνα να δουλέψουν, για την Αγγλική καμπίνα συγγνώμη, να δουλέψει και λίγο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή σα για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου και να ευχαριστήσω τους παρόντες. Σας έδωσα τη δομή της ομιλίας μου. Ε, θα περιοριστώ στο τέταρτο. Η πρόταση περιέχει λίγες αλλαγές σε σχέση με την κοινή οργάνωση αγοράς. Μερικές αλλαγές είναι πραγματικά ευπρόσδεκτες. Οι κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, η βελτίωση και απλούστευση των κανόνων για τις γεωγραφικές ενδείξεις είναι ένα θετικό στοιχείο της νέας πρότασης. Επίσης, η διατήρηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων σε, το σε τομείς όπως ο αμπελοϊνικός είναι άλλο θετικό στοιχείο. Η η διατήρηση του προϋπολογισμού για τα οποροκυπευτικά επιχειρησιακά προγράμματα χωρίς δημοσιονομικό προϋπολογισμό, χωρίς δημοσιονομικό περιορισμό. Αυτό είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο. Πιθανότητα ε, επέκταση της χρηματοδότησης των επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων και σε άλλους τομείς. Επίσης ε, θετικό στοιχείο. Λίγε πάντως είναι οι αλλαγές, γιατί με τον κανονισμό Omnibus περιλήφθηκαν κάποιες θετικέ καινοτομίε, χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διαδραμάτισε εκεί σημαντικό ρόλο και θετι... οι θετικέ εξελίξει ενισχύθηκαν από την πρόσφατη νομολογία του 10 για τα ραδίκια Αντίβ. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα ε, στην ακρόαση που είχαμε μιλήσαμε για αυτό το θέμα της νομολογίας ε, του ΔΕΚ για την περίπτωση των γαλλικών ραδικιών αντίβ και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την ε, απόφαση και την υπεροχή της Γεωργίας έναντι των κανόνων ανταγωνισμού. Αυτά και θα εψέλθω άμεσα στις 28 προτάσεις που θα σας κάνω και τις συστάσεις που ελπίζω να σας χρησιμεύσουν. Οχτώ από αυτές δεν αφορούν την ε, κανονιστική ρύθμιση, αλλά είναι σημαντικές και 21 από τις 29 προτάσεις αφορούν τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Καταρχήν, είμαι υπέρ του αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα πολιετέ αποθεματικό κρίση. Και αυτό το ζήτημα το έχετε επανειλημμένο συζητήσει. Μια και οι κρίσει είναι απρόβλεπτε, το αποθεματικό για τι κρίσει είναι απαραίτητο και με πολιετή χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, ήδη έχετε εγκρίνει την πρόταση ε, του κυρίου Δεκάστρο και τη σχετική γνωμοδότηση. Είναι κέριο αυτό το σημείο αν θέλουμε πραγματικά βελτίωση του γεωργικού εισοδήματο. Ε, του, του πρώτου κρίκου της ε, διατροφικής αλυσίδας. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ε, ζήτησε να στηρίξουμε τις τοπικές αγορές, τη βραχή αλυσίδα εφοδιασμού και ήδη εδώ και καιρό στηρίζεται τη πολιτική ποιότητα με τις ονομασίες προέλευσης, την βιολογική γεωργία, τις περιβαλλοντικές πρακτικές, οτιδήποτε δηλαδή χρησιμεύει για τη διαφοροποίηση των κινδύνων εντός τη αγροτική εκμετάλλευση. Και γι' αυτό οι τοπικές αγορές και οι βραχές αλυσίδες ενεφοδιασμού είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Επίσης, προληπτική εξοικονόμηση. Βέβαια, αυτό είναι αμυγό εθνική αρμοδιότητα, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το λέει και η Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη. Αυτή η, προληπτική εξοικονόμηση είναι πολύ σημαντική και σε κάποιες χώρες ε, σίγουρα η φορολογία ε, είναι πιο φιλική προς επενδύσεις παρά προς τη, στην αποταμίευση, αλλά εδώ θα έλεγα να προτείνουμε κάποια ενάψματα και για την ε, προληπτική αποταμίευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε και την αιρεσιμότητα και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διαφοροποίησης και άλλο θετικό επίσης ε, στοιχείο που θα πρέπει να στηρίξουμε από τη νέα πρόταση. Ένα θέμα που παραλείπεται από τις προτάσεις, παρόλο που κατά τη γνώμη μου έχει σημασία, είναι ότι στα αποτελέσματα των πλεονεκτημάτων που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνεται στους δικαιούχους, ε, περιλαμβάνονται στους δικαιούχους και οι εμπορικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που έχουν ε, ε, επαρκή τζίρο ώστε να μπορούν να εξισορροπούν το σχετισμό δυνάμεων στην αλυσίδα, στην διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή θα πρέπει να τιμωρούμε τους πετυχημένους παραγωγούς που δεν εμπίπτουν πια στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι περιλαμβάνουμε και τις εμπορικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κάποια επιχειρηματικά κεφάλαια από τον πρώτο πυλώνα σε επίπεδο 3%. Κατά τη γνώμη μου θα είχε νόημα να συγχωνεύσουμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις με τις ε, ενισχύσεις από αυτό το επιχειρησιακό σύστημα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε συνδεδεμένη ενίσχυση για τον ίνο, κάποια ευρώ ε, για το πρόβιο κρέας, ε, μερικά ευρώ ανακεφάλι αλλά θα μπορούσαμε μία στήριξη να δώσουμε σε διεπαγγελματική οργάνωση, σε οργάνωση παραγωγών ή ενώση οργάνωση παραγωγών για να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν καλύτερα. Η στήριξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις οργανώσεις παραγωγών θα έλεγα να συγχωνευτούν με τις συνδεδεμένε συνδεδεμένες ενισχύσεις και με την αύξηση αυτού του 3% και σε επίπεδο ελέγχου θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επιθεωρητές, οι ελεκτές να μην δίνανται ε, να επιβάλλουν αναδρομικά τα αποτελέσματα των ελέγχων τους πριν, να ανάγονται δηλαδή σε 4-5 χρόνια πριν, γιατί κάτι έτσι θα ήταν πολύ περίπλοκο. Τώρα επισέρχομαι στον κανονισμό καθ' αυτό. Τέσσερις είναι οι βασικές αρχές κατά τη γνώμη μου στις δύσκολες δημοσιονομικές ε, περιόδους θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σε όσα ε, έχουν θετικό αντίκτυπο στο γεωρικό εισόδημα και στην ευημερία του καταναλωτή. Και ε, μάλιστα δεν έχουν και δημοσιονομικό αντίκτυπο. Θα πρέπει λοιπόν στο βασικό κανονισμό να αφήσουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές Είπαμε την ομολογία του ΔΕΚ για τα ραδίκια αντίφ. Να αφήσουμε όλε τι δυνατέ λύσει ώστε οι γεωργοί να μπορούν να χρησιμοποιούν όλε αυτέ τι πιθανότητε, δυνατότητε, αν το κρίνουν σκόπιμο. Να αφήσουμε λοιπόν ένα ευρύτατο φάσμα δυνατοτήτων και μηχανισμών που εμπίπτουν στην κοινή γεωργική πολιτική και που υπερέχουν σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού οι γεωργοί θα εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα, αλλά να έχουν δυνατότητα να επιλέξουν από ένα ευρύτατο φάσμα μέτρων και μηχανισμών. Και αυτέ οι δυνατότητε, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο κείμενο του κανονισμού. Εξού και οι δικέ μου συστάσεις και προτάσει. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τη αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαφάνεια τη αγορά. Ήδη έχουμε τέσσερα τομεακά παρατηρητήρια, έχουμε και τον πίνακα επιδόσεων αποτελεσμάτων μάλλον που εκδίδεται τακτικά. Θα ζητούσαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των γεωργικών αγορών για να έχουμε πιο συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες ε, για όλους σε ό,τι αφορά τους ε, τομείς που καλύπτονται. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη για τους συνεταιρισμούς. Χρειάζονται και άλλες μελέτες και άλλες πληροφορίες για τα στατιστικά στοιχεία που έχει το σύνολο του κλάδου τη διατροφική αλυσίδα. Και θα πρέπει επίση να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων για του συνεταιρισμού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε στατιστικέ ε, πληροφορίε και για τα βιολογικά προϊόντα. Και τακτικά, περιοδικά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιστά έκθεση για την πρόοδο που επιτυχάνεται σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια τη αγορά. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια παρέμβαση, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γεωργικών Αγορών, και σε ό,τι φορά τις μελέτες, θα θέλαμε ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, ώστε με βάση τακτικές εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εντοπίζονται τα προβλήματα που ενδεχομένω θα ε, επηρεάσουν τις αγορές. Στο παρόν σύστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δύναται να παρεμβεί την κατάλληλη στιγμή και όταν το κρίνει σκόπιμο. Αλλά πώς θα γίνεται σωστή διαχείριση ε, κινδύνων με τέτοια βεβαιότητα. Γι' αυτό, πριν από 12 χρόνια, στην έκθεση παραχή που είχαμε επιβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαχείριση κινδύνου, ζητήσαμε σαφέστατα κριτήρια δημόσια παρέμβαση. Θα πρέπει εκ των προτέρων να είναι γνωστό πότε και τι ακριβώ δικαιούται να κάνει η διοίκηση. Και μάλιστα πολλοί ευρωβουλευτέ ζήτησαν από την Επιτροπή να παρέμβει στην αγορά ζάχαρης Υπήρξε όμω ε, μια πολύ μεγάλη φαιά ζώνη, μια μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτή την αβεβαιότητα θα πρέπει να την περιορίσουμε και να γνωρίζουμε πότε θα γίνεται μια δημόσια παρέμβαση στι αγορές και θα πρέπει και οι οικονομικοί τελεστέ να μπορούν να διαχειριστούν του κινδύνου όπω θέλουν. Θα πρέπει όμω να υπάρχει προβλεψιμότητα και βεβαιότητα. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι τιμέ αναφορά, όπω λέγονται τώρα, στον, στον τομέα. Μερικοί ζήτησαν αύξηση των τιμών αναφορά. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά σε πρόσφατη μελέτη για το γάλα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του γάλακτο στο σκόνη και να αυξηθεί η τιμή του νοπού γάλακτο και του βουτύρου. Γιατί έχουμε κάποιε τιμέ που αφορούν το παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν η δημόσια παρέμβαση να παραμένει ως δίκτυο ασφάλεια αλλά να ενεργοποιείται ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά. Και μάλιστα όταν χρειάστηκε παρέμβαση στην αγορά προκυπευτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αύξησε τις τιμές απόσυρσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών. Αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Νταντά στην ε, σχετική έκθεση και η νομολογία το επιβεβαίωσε θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό των εμπορικών ε, οργανώσεων παραγωγών που είναι επιχειρήσεις που καλύπτονται πλήρως όπως είπα προηγουμένως και με το απέδειξε και το δικαστήριο με την ομολογία για τα λαδί και αντίφ από τις υπόλοιπες ομάδες διαπραγμάτευσης που είναι πολύ χρήσιμες οντότητες και μάλιστα Είχαμε ένα εξαιρετικό σεμινάριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δόθηκαν παραδείγματα θαυμάσια από την αγορά ε, βόηου κρέατος ε, και από το τομέα γάλακτος. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, άλλε οντότητε. Δεν καλύπτονται από την ομολογία για τα ραδίκια αντίβ. Δεν είναι δηλαδή οι εμπορικέ οργανώσει παραγωγών. Οπότε, καλύπτονται μόνο οι εμπορικέ οργανώσει παραγωγών και οι ενώσει οργανώσει παραγωγών που θα μπορούν να δικαιούνται να προσαρμόσουν σε ποιότητα και ποσότητα την προσφορά στη ζήτηση, χωρίς προηγούμενη άδεια, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις, στα απορροκυπευτικά, οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να, αποσύρουν όποτε θέλουν και ό,τι θέλουν, χωρίς άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η, το νόημα του, άρθρου 152 και των εδαφείων του. Επίσης, μία επιχείρηση μπορεί να ορίσει τις τιμές όπως επιθυμεί και μία εμπορική οργάνωση παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορεί κάλλιστα να έχει τη δική του πολιτική για τις τιμές και αν αποφασίσει να μην πουλήσει σε συγκεκριμένη τιμή θα πρέπει να έχει την ελευθερία να το κάνει. Επίσης, θα πρέπει να διευκολύνουμε την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση του για τους νέους τομείς να αποφύγω μια χρονοβόρα διαδικασία αναγνώρισης. Θα μπορούσε και να επεκταθεί το θέμα των σημερινών συνεταιρισμών και να δώσουμε τα διεπιστευτήριά τους στις οργανώσεις παραγωγών και σε ενός οργανώσεων παραγωγών. Και επαναλαμβάνω, επικεντρώνουμε στις εμπορικές οργανώσεις παραγωγών και ενός οργανώσεων παραγωγών. Τα υπόλοιπα είναι ομάδες διαπραγμάτευση. και για τις διασυνοριακές οργανώσεις και ενός οργανώσεων παραγωγών υπάρχουν στον κανονισμό αλλά δεν προβλέπονται ξεχωριστά. Στην Ισπανία οι οργανώσεις παραγωγών είναι κυρίως περιφερειακές. Όταν όμως έχουν μέλη σε διάφορες περιφέρειες, η εποπτεία ασκείται από την κεντρική κυβέρνηση. Μία διασυνοριακή οργάνωση παραγωγών προϋποθέτει συνεργασία διαφόρων παραγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταλήξουμε στην Ευρώπη τη πραγματικότητα και στην Ευρώπη των επιχειρήσεων. Αυτέ οι διασυνοριακέ οργανώσει παραγωγών σήμερα είναι ο εφιάλτη των εθνικών διηγήσεων που, θα, που καλούνται να τι διαχειριστούν. Γι' αυτό λοιπόν οι οργανώσει παραγωγών, κυρίω οι διασυνοριακέ θα πρέπει να ε, εμπίπτουν στο, στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως στην Ισπανία οι διαπεριφερειακές οργανώσεις παραγωγών ε, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ε, κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, ό,τι αφορά τη, συνεργασία μεταξύ περιφερειών και κρατών για τις οργανώσεις παραγωγών ή ενός οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να προτείνεται να προβλέπεται η δυνατότητα διασυνοριακής συνεργασίας. Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ε, δημιουργούνται με πρωτοβουλία των οργανώσεων παραγωγών. Εγώ προτείνω να γίνονται με πρωτοβουλία και άλλων ενώσεων παραγωγών, ε, οργανώσεων παραγωγών, όχι μόνο από, μετά από πρωτοβουλία οργανώσεων παραγωγών, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό. Επίσης, όπως προβλέψαμε τη δυνατότητα της Ένωσης Οργάνωσης Παραγωγών, να προβλέψουμε και την οντότητα της Ένωσης Διαπαγγελματικών Οργανώσεων. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο ώστε και στη, να υπάρχει και Ένωση Διαπαγγελματικών Οργανώσεων που να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που τις εκχωρεί η Διαπαγγελματική οργάνωση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Υποβάλλω λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις ε, και πιστεύω ότι όταν είμαστε ουδέτεροι δημοσιονομικά μπορούμε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Επίσης, σε ένα βιβλίο του Παόλου Ντεκάστρο που φεύγει, αλλά το βιβλίο του μένει, το βιβλίο του μένει. Ο κύριος Δεκάστρο λοιπόν είπε ότι η ιδιωτική παρέμβαση και η ιδιωτική διαχείριση ε, της κρίσης είναι ένα καθυσυχαστικός μηχανισμός για την αγορά η ιδιωτική παρέμβαση μόνο προληπτικά έχει νόημα. Όχι λοιπόν θα πρέπει να έχει λάβει προ... προκατακτική άδεια, αλλά θα πρέπει να στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβαση. Όταν αρχίζει η πυρκαγιά, τότε οι διαπαγγελματικέ οργανώσει, οι οργανώσει παραγών και οι ενώσει οργανώσει παραγωγών μπορούν να συμβάλλουν για να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι προκαταρκτικές ε, ενέργειες θα πρέπει να στηριχθούν. Τώρα, οι διαπαγγελματικέ οργανώσεις επίσης θα, μπορούν, θα πρέπει να μπορούν να επεμβαίνουν στη διαχείριση των κρίσεων και των αγορών. Αυτή τη στιγμή προβλέπονται μόνο για τις διαπαγγελματικές οργανώσεις σε κάποιες ονομασίες προέλευσης ε, τυριών και άλλων προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε το φάσμα ώστε να είναι δυνατή η χρήση του μηχανισμού για τομεί που θέλουν ποιοτικά ή άλλα προϊόντα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο των διαπαγγελματικών οργανώσεων οι ανώσει οργανώσεων παραγωγών και οι διασυνοριακέ ενώσει οργανώσεων παραγωγών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ω συνδεδεμένα μέλη και οργανώσει παραγωγών, διαπαγγελματικέ οργανώσει ενό οργανώσεων παραγωγών και τρίτων χωρών εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και το τελευταίο στοιχείο. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά θα πρέπει να διευρύνουμε την νομική, το, νομικό πεδίο του κανονισμού και σε διατάξεις που ε, ε εγκρίνουν οι οργανώσεις παραγωγών ενός οργανώσεων παραγωγών ε, για τους ε, γεωργούς, ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στους ε, εισηγητές μας. Θα μιλήσουν ο κύριος Ερντός, η κυρία Γιλέρα, Σένρα, Σάντος. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο στη συζήτηση, Φλάναγκαν, Καλινόφσκι. Καλύτερα να το ξέρω από τώρα για να κατανείμω το χρόνο. Α, κύριε Ρομπέρτο, φαντάστηκα ότι θα ζητήσετε και εσείς τον λόγο. Δύο με τρία λεπτό καθένας, παρακαλώ. Ο κύριος Έρντος. Μετά από δύο λεπτά διακριτικά θα αρχίσω να σηκώνω το σφυράκι. Ε, jelenlévő Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο πτυχές και δύο ερωτήσεις δηλαδή προς τους εμπειρογνώμονες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το νέο μοντέλο απόδοσης ε, Ε, κινδυνεύει λόγω των προϋποθέσεων και της χρήσης των άμεσων, των άμεσων πληρωμών. Ε, ε, αυτά που προτείνονται δεν είναι σύμφωνα με τις συνθήκες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει ποιοι γεωργοί μπορούν να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές και ποιοι όχι και ποιες, ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν. Γιατί αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της γεωργικής μας πολιτικής εμπίπτυσης, αρμοδιότητες δηλαδή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γι' αυτό θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Καταρχάς, πώς βλέπουν το θέμα αυτό από την νομική άποψη και δεύτερον, από την άποψη των γεωργών, τι πιστεύουν. Δεύτερη παρατήρηση. Το ερώτημα που σχετίζεται με την εσωτερική σύγκληση των κρατών μελών και την απέτηση σύγκληση, δεν θα είναι σωστό να επικρατήσει αυτό το, το αυτός ο στόχος ε, εις βάρος άλλων γεωργών αλλού στην Ένωση. Είναι άδικο για να υπάρξει εξωτερική σύγκληση να συνεχιστεί η στήριξη κρατών όπως η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι περιοτείνετε εσείς για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των τριών εμπειρογνωμόνων και πολύ ε, πρακτική. Η πρώτη παρέμβαση είναι το κατά πόσο με βάση τα αποτελέσματα η Κομισιόν να, μπορεί να προσθέσει νομιμότητα σε αυτή την πολιτική. Μπορείτε αυτό να μου το εξηγήσετε, είναι δυνατό, είναι πιθανό, αλλά αυτό το, το, θεμητό χαρακτήρα, το νόμιμο, το νόμιμο χαρακτήρα που λέτε, πώς ακριβώς θα αυξηθεί η νομιμότητα. Ε, απλοποίηση, απλοποίηση, απλούστευση στην Κομισιόν, ναι, και στα κρατημέλη, γιατί μπορεί να αλλάξουμε ρόλους ένα πρόβλημα με ένα άλλο, ένα κατόχλη με ένα άλλο. Δηλαδή, αντί να έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε την ε, κυβέρνηση της Ισπανίας. Ε, δεν ξέρω. Και έπειτα εσωτερική αγορά και διαφορετική εφαρμογή που ε, φέρνει αυτό το πρότυπο με βάση τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι υπέρ του κάπινγκ. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχουν και ηθικά θέματα. Οι δημόσιες ε, ε, ενισχύσεις θα πρέπει να μετρώνται σαφώς και να ξέρουμε πού πάνε. Εγώ το λέω για στη δική μου περιφέρεια. Έχουμε ε, εκμεταλλεύσεις με 50.000, 500.000 ε, ευρώ. Είναι ένα ε, θέμα ότι έστω και συμβολικά θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο και έπειτα για την εφαρμογή της απασχόλησης από τις 60.000 στις 100.000 ευρώ για μένα δεν είναι σωστό να προσαρμόζουμε ανά θέση επασχόλησης που μπορεί να επιδοτηθεί. Αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο, γιατί υπάρχουν χώρες όπως η δική μου που είναι μεγάλες εκμεταλλεύσεις και πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι, ένα ανώτατο όριο μάλλον. Τώρα, το θέμα των ε, κοινωνικών ε, ε, συνεισφορών και το τελευταίο εκεί που λέτε ε, οι οργανώσεις της ΕΚΟΑ νομίζω πως κατευθύνεται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε ένα τομέα και γι' αυτό θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς ε, θα αποφασίσουμε όταν λέτε ότι πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης. Όμως ε, Πώς θα αποφασίζει η Κομισιόν με με σε τι αντιστοιχεί το γεγονός ότι μια επιχείρηση με μόνο εμπορικό χαρακτήρα θα περιλαμβάνει στους εταίρους μια, μια μεγάλη οργάνωση παραγωγών. Ενώ ο, ο κάτοχος είναι ο αρχηγός, όπως λέμε δηλαδή, τι θα βάλουμε το λίκο να τα πρόβατα, όπως λέμε εμείς στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χόιμπουχ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναρπαστικές ήταν οι παρουσιάσεις. Επιβεβαιώθηκαν πολλά από τα όσα ήδη φοβόμουν ε, και το είπατε όλοι πάνω κάτω αυτό. Ότι είναι καλές οι προθέσεις, αλλά πάρα πολύ αδύναμη διατύπωση. Ε, δεν είμαστε αρκετά ακριβείς Επίσης είπατε ότι πολλές φορές υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων και δυνατοτήτων στα κράτη-μέλη. Και από αυτό και μόνο το λόγο τελικά θα πρέπει να υπολογίζουμε σε διαφορετική εφαρμογή ανά χώρα. Όλες αυτές λοιπόν οι αγωνίες μου επιβεβαιώθηκαν και που οδηγούμαστε σε συνολική αποδυνάμωση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κάτι όπως, όμως που μου λείπει και αυτό μου το επιβεβαιώσατε είναι οι ποσοτικές ε, ε, ρυθμίσεις. Ε, ότι τόσα θα πρέπει να πηγαίνουν για τα κοινωνικά, τόσα θα πρέπει να πηγαίνουν για τα περιβαλλοντικά και εκεί είναι θολό το τοπίο. Και είναι τόσο διαφορετική η στόχη μεταξύ τους, οικονομική, κοινωνική, οικολογική που καμιά φορά μπορεί να είναι και αντιφατική. Διότι δεν έχουμε σταθμίσει κάθε φορά ε, τις ε, καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη-μέλη, τις ανάγκες και τις ε, προτιμήσεις τους. Άκουσα επίσης να συμφωνείτε σε πολλά από αυτά που με απασχολούν. Αυτά τα eco-schemes, τα οικολογικά σχήματα που αφορούν και τους δύο πυλώνες και τον πρώτο πυλώνα δηλαδή. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα μειωθεί τώρα η γραφειοκρατία αν βάλουμε τέτοια οικολογικά σχήματα και στον πρώτο πυλώνα, που είναι προγράμματα αντίστοιχα με του δευτέρου πυλώνα. Με αντίστοιχους μηχανισμούς δηλαδή. Ποιος έχει πρόσβαση, ποιος έχει δικαίωμα, πώς ελέγχεται, πώς εφαρμόζεται. Και στους δύο πυλώνες δηλαδή θα έχουμε διαφορετικές προσφορές ε, με υπερβολική γραφειοκρατία ε, στα αγροκτήματα και στις εκμεταλλεύσεις και ποιος θα τα βγάζει πέρα. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πολλές προσφορές για το κλίμα, για το περιβάλλον και για τα κοινωνικά, αλλά δεν έχει νόημα να αφήνουμε να επικρατεί τέτοια βεβαιότητα και τέτοια ανισότητα και να το αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν θα έχουμε κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί τελικά όλοι πουλάμε στην ίδια εσωτερική αγορά και εγώ αγρότησα είμαι. Και αν δεν είναι οι ίδιοι κανόνες του ανταγωνισμού έχω μεγάλο πρόβλημα. Ε, διαχείριση των κρίσεων ε, των αγορών. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και υπολείπεται η πρόταση κατά πολύ. Δεν νομίζω ότι λύνεται αυτό με ε, ασφάλειες όταν καταραίουν οι αγορές. Τι να ασφαλίσεις. Το βασικό εισόδημα, πέρα από τις ενισχύσεις και τις πληρωμές, ε, είναι το εισόδημα που έχει ε, κάποιος από την πώληση ε, του προϊόντος που παράγει. Αυτή είναι η έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης. Και μια τελευταία παρατήρηση για την οροφή, το κάπινγκ, κινδυνεύει να ξεδοντιαστεί. Εάν μπορούμε να εκπίπτουμε κάθε ε, κόστος μισολογικό ακόμα και το εικονικό κόστος που θα ε, αφορούσε τους μισθούς της οικογένειας που δεν πληρώνονται. Μα εγώ για να προσλάβω κάποιο στο αγρόκτημα θα πρέπει να το χρειάζομαι στην επιχείρηση, στην εκμετάλλευση και όχι να το παίρνω για να παίρνω την επιδότηση. Δηλαδή να παράγει ο άνθρωπος κάτι, να παράγει αξία και οικονομική αξία χρειάζεται τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που έχουμε πάρει. Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες μας γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες που μας έκαναν και πολύ χρήσιμες οι συστάσεις τους. Εγώ θα σταθώ στην ανάγκη της μείωση της γραφειοκρατίας που ταλανίζει τους ε, παραγωγούς. Θέλουμε να πλουστεύσουμε το περίπλοκο πλέγμα κανονισμών της ΚΑΠ και αυτός ήταν ένας από τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ειδικής μας Επιτροπής και των, των μελών της. Πιστεύουμε ότι οι οργανώσεις παραγών θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Δηλαδή να επικεντρωθούν στον κοινωνικο-οικονομικό τους ρόλο και να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ασφάλειας. Και γι' αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η γραφειοκρατία να μην είναι ένα βάρος που θα πρέπει να ε, κουβαλάνε οι γεωργοί ε, και ένα είδος εξηλαίωσης για τις ενισχύσεις που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη τώρα καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχου και διαχείρισης των σχέσεων με τις οργανώσεις παραγωγών. Χρειάζεται ε, μια μεγαλύτερη ελαστικότητα και αυτή είναι ευπρόσδεκτη αλλαγή και τα κράτη-μέλη θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν στο επίπεδό τους τις απαραίτητες προσπάθειες. Βέβαια, μιλάμε για κοινή γεωρική πολιτική. Γι' αυτό θα πρέπει τα αποτελέσματα και έλεγχοι να είναι σε τελικό βαθμό αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα πρέπει κατά ανάγκη να σκεφτούμε τι γίνεται με τις οργανώσεις παραγωγών. Και μάλιστα από την ανάλυση σας ε, κατάλαβα ότι η έμπρακτη εφαρμογή αυτού του νέου delivery model, του μοντέλου παροχής αποτελεσμάτων, θα αυξήσει αισθητά την περιπλοκότητα και το γραφειοκρατικό άχθος για τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Εσείς τι άποψη έχετε. Κατά τη γνώμη σας, ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού του νέου delivery model. Πώς θα επηρεάσει αυτό το νέο μοντέλο παροχής παροχή αποτελεσμάτων, τη γραφειοκρατία και πώς θα επιβαρύνει, ε, θα επιβαρύνει περαιτέρω τους ε, παραγωγούς, τους γεωργού. Ευχαριστώ. Κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους τρει καλεσμένους μας για τις ε, παρουσιάσεις τους και να κάνω μια ερώτηση που την απευθύνω και στους τρεις. Εδώ και πολύ καιρό μιλούμε και από εδώ που είμαι μέλος της Επιτροπής Άγκρη αλλά και σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για τις κρίσεις που διανύουμε η παραγωγή του γεωργικού κλάδου. Μιλούμε για τις δυσκολίες που έχουν οι γεωργοί, για την απροθυμία των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργική δραστηριότητα, για την γύραση του αγροτικού πληθυσμού, για την απερίμωση των αγροτικών ζωνών και της υπαίθρου. Και νομίζω ότι την ουσία έχουμε ένα βασικό πρόβλημα με τις τιμές ή με το γεωργικό εισόδημα, με την ανταμοιβή τους δηλαδή για, το, για τη γεωργική τους δραστηριότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ερωτώ λοιπόν, μήπως πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε και πάλι δημόσιες πολιτικές αποφασιστικές και οι τιμές παραγωγού να βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο της νέας ΚΑΠ και να είναι δίκαιες και μέσω δημόσιων πολιτικών να έχουμε μηχανισμούς ε, ρύθμισης ε, της παραγωγής της αγορές. Ο πρώτος καλεσμένος μίλησε για ε, περιβαλλοντικούς δείκτες που δεν συνδέονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Τι δείκτες ε, εννοείστε και πώς μπορούν να συμβάλλουν οι δείκτες αυτοί για, τη... για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Τι δείκτες ακριβώς εννοούσατε όταν είπατε για δείκτε που δεν εμπίπτουν στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίση, μιλήσατε για διαβουλεύσει και για κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Μιλήσατε για την κοινή λήψη αποφάσεων, για τη συναπόφαση. Κατά τη γνώμη σα, τι ρόλο θα πρέπει να έχουν οι οργανώσεις αγροτών, όχι οι οργανώσεις παραγωγών, οι αγροτικές οργανώσεις, τι ρόλο θα μπορούσαν να έχουν στη λήψη αποφάσεων, γιατί και αυτές θα πρέπει ε, να λάβουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Οι αγροτικές οργανώσεις και ενώσεις. Επίσης, ε, δεύτερος καλεσμένος μας μίλησε για την ισχυρή εξάρτηση του εισοδήματος από τις δημόσιες ενισχύσεις, τις, ενισχύσεις, ε, τις γεωργικές ενισχύσεις. Και είπε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ναι, όντως, θα πρέπει να μειωθεί η συμβολή των άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα, να είναι υψηλότερε σε τιμέ και να ανταμείβουν οι τιμέ ε, των γεωργών. Αλλά και το θέμα το μέγεθο ε, των γεωρικών εκμεταλλεύσεων είναι σημαντικό. Είπατε ότι υπάρχουν πολύ μικρέ ε, γεωρικές εκμεταλλεύσεις, υπερβολικά μικρέ. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το ιδανικό μέγεθο μια γεωρικής εκμετάλλευση. Εδώ και 30 χρόνια ακούω την εποδό θα πρέπει να αυξήσουμε το μέγεθο των γεωρικών εκμεταλλεύσεων. Βέβαια, προ τα κάτω δεν υπάρχει όριο, γιατί όταν αφανίζονται οι μικρέ εκμεταλλεύσει, οι επόμενες είναι και πάλι μικρές. Ποιο είναι κατά τη γνώμη το ιδεώδες μέγεθος για μια αγιορική εκμετάλλευση και πιστεύετε ότι θα πρέπει να επέμβουμε σε επίπεδο τιμών για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Κύριε Αθκάρατε, θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λίγο αυτό που είπατε για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των οργανώσεων ε, παραγωγών ώστε τα μέτρα τους να εφαρμόζονται στους παραγωγούς. Γιατί δεν κατάλαβα ακριβώ αυτό που είπατε. Τώρα, ποιο είναι το ιδεώδες μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης. Τι να σας πω, εξαρτάται από τις συνθήκες. Ο κύριος Καλινόφσκι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν ήμουν από την αρχή στη συνεδρίαση και έχασα ένα τμήμα των παρεμβάσεων. Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και απευθύνω τι τις παρατηρήσεις μου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εξή. Έχουμε τις άμεσες ενισχύσεις που είναι ανακατεμικές, ανακατανεμητικές. Εγώ είμαι υπέρ αυτού του, του μηχανισμού, αλλά θα πρέπει αυτό το μηχανισμό να το συνδυάσουμε με τα άρθρα 4 και 16 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που λένε ότι τα κράτη-μέλη στα στρατηγικά του σχέδια θα πρέπει να προσδιορίσουν την έννοια του ενεργού αγρότη. Το αγρότη που ασκεί πραγματικά γεωρική δραστηριότητα. Και θα πρέπει όμως να ελέγξουμε αυτό τον ορισμό. Γιατί ο ορισμός ε, θα πρέπει να έχει ένα νόημα και να μην πηγαίνουν ε, κοινοτικά κονδύλια σε μη γεωργούς. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την, από την Πολωνία. Ε, ένα εκατομμύριο τριακόσι χιλιάδες ε, στην Πολωνία υποβάλλουν αιτήματα για άμεσες ενισχύσεις. Αλλά από αυτό το 1.300.000 μόνο μερικές χιλιάδες είναι οι πραγματικά ενεργοί γεωργοί, δηλαδή αυτοί που πραγματικά ασκούν γεωργική δραστηριότητα. Οι υπόλοιπε 700.000 είναι ε, ιδιοκτήτες ε, μερικών δεκάδων ε, εκταρίων που δεν ασκούν μόνο τη συγκεκριτική δραστηριότητα αλλά εκμισθώνουν τα χωράφια τους. Επίσης έχουμε έναν γεωργό που έχει 80 εκτάρια. Τα 40 είναι δικά του και για αυτά τα εκτάρια υποβάλλει αίτηση και τα υπόλοιπα 40 εκτάρια τα δίνει στον ε, ιδιοκτήτη από την αγρομίσθωση που έχει. Ποιος κάνει την, ε, τον έλεγχο και δεν έχει και ε, φιλο, οικολογικοποίηση. Το πρασίνισμα δεν το εφαρμόζει, ενώ ο πραγματικός γερός είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Επίσης, επειδή κάνει για περιορισμένο χωράφι το, την, το, την αίτησή του, δεν μπορεί να λάβει ενισχύσει για τα μηχανήματα για το σύνολο της έκτασης ή δεν μπορεί να λάβει την επιδότηση για τα γεωρικά καύσιμα. Επίσης, ακόμη και για τις αποζημιώσεις που ζητούν για την ξηρασία. Δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για το σύνολο των εκταρίων που καλλιεργούν, αλλά μόνο για το δικό του τμήμα και όχι για αυτό που μεταφέρουν στον ε, πραγματικό ιδιοκτήτη. Οπότε ο ορισμός του ενεργού αγρότη θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμος, ελέγξιμος, γιατί αν δεν καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο και πάλι θα είναι όλα θεωρητικά και πάλι θα μπορούμε να μιλούμε για να μοποιήσει αυτού του μηχανισμού της γεωργικής πολιτικής. Ε, κάπως μπερδεμένα μας τα είπε, ούτε εγώ δεν τα κατάλαβα όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζροπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για τη διοργάνωση του σεμιναρίου τούτου. Είναι πολύ καλό να ακούμε εδώ επιστήμονες, εμπειρογνώμονες που έχουν ασχοληθεί ε, με ε, το νομοθέτημα που καλούμαστε εμείς να ε, ψηφίσουμε για να αποφασίσουμε με τα λόγου γνώσεων. χρειάζεται απλούστευση, όπως και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και στην κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό λυπάμαι λίγο που στην πρόταση που έχουμε για τη σύγκληση ε, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. 75% του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι μια πρόταση ενδεκτική μόνο, προσανατολιστική. Στο παρελθόν λέγαμε ότι μέχρι το 2013 θα πρέπει να έχουμε επιτύχει τη σύγκληση ε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Καμία σχέση. Και πέντε χρόνια μετά ούτε στο 75% δεν έχουμε φτάσει και έχουμε επεμπολίσει το 100%, τώρα μιλάμε για 75%, ε, είναι εις βάρος των αγροτών των αλλητολικών χωρών και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αυτό πριν από μια πενταετία. Θα πάνε όλα στο βρόντο αυτά, όλες οι προσπάθειες, εάν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε την απερίμωση της υπαίθρου με την αστιφιλία, με τη διαρροή ε, των ε, εγκεφάλων και με την πίεση που υφίστανται όλες αυτές οι περιφέρειες. Αλλιώς πραγματικά δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Φεύγει η γνώση, η καινοτομία, ε, ε, οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ποιος θα κληθεί να τα εφαρμόσει όλα αυτά τα ωραία που προτείνονται. όσο ε, καλή και ωραία και να είναι η κοινή γεωργική πολιτική, δεν βοηθάει αν δεν υπάρχει κάποιο να την εφαρμόσει, να την υλοποιήσει επιτόπου και να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν από τα κέρδη των προϊόντων που παράγουν. Αλλιώς πραγματικά όλα αυτά πάνε στον βρόντο. Γερνάνε οι αγρότες, οι νέοι δεν εγκαθίστανται στην Ήπεθρο. Και υπάρχουν και πολλοί πενιντάριδες που δεν βλέπουν καμία προοπτική για την εκμετάλλευσή τους. Όλα αυτά τα ξέρουν οι αγρότες, τα βλέπουν. Και όποιος δουλεύει στη Γεωργία παίρνει το μισό μισθό από το βιομηχανικό εργάτη. Γιατί να πάει να γίνει αγροτικός εργάτης. Έχουμε φιλόδοξους στόχους και ευγενείς για τα τρόφιμα, για την ποιότητα κτλ. Και πριν από δύο χρόνια δεν είχαμε βούτυρο στην Ευρώπη. Τι να την κάνουμε αυτή τη νέα πολιτική μέχρι το 2027 ε, για τα ποιοτικά και καλά προϊόντα. Αν δεν συζητήσουμε ε, για ε, το πώς θα εξασφαλίσουμε τα βασικά για τον πληθυσμό και όχι τις εξαγωγές και, την υψηλή μεταποίηση, τα βασικά καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Επίσης, σε κάποια κράτη-μέλη, με αυτά τα οικολογικά τώρα σχήματα και προγράμματα, υπάρχει πρόβλημα. Διότι η επιδότηση δεν είναι ίδια. Οι άλλες χώρες δίνουν 50% και άλλες 150% για την ίδια υπηρεσία. Δεν μπορεί ένας Πολωνός αγρότης να παίρνουν πολύ λιγότερα από κράτη-μέλη και λιγότερα οι βαλτικές χώρες δίνουν και ακόμα λιγότερα παίρνει ο Βούλγαρος αγρότης. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον Ανατολή Δύση θα πρέπει να έχει ε, την ίδια μεταχείριση που δεν έγινε πριν την ένταξη. Είναι δύσκολη η κατάσταση και και παντού. Κυρίε και κύριοι, εξελίσσαμε το κατάλογο των αγορητών από την Επιτροπή. Ε, δεν καλωσόρισα πριν και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. Μέγκελε. Πριν όμως δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δώσω στον κύριο Φλάναγκαν. right, no problem. Ε, ναι, πολύ ωραία, κάνα πρόβλημα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Έχω μια ερώτηση συγκεκριμένα για τον κύριο, το δεύτερο που πήρε το λόγο. Είπατε ότι οι ενισχύσεις οδηγούν σε ανισότητες και πώς η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα το καλύψει αυτό. Εγώ συμφωνώ με την εξήγηση του Άλεν Μάθιους που λέει ότι δεν, έχουν, δεν έχει νόημα ε, όλο αυτό. Ήλπιζα ερχόμενος εδώ ότι θα βλέπαμε μια σωστή ανακατανομή και ότι θα απομακρυνόμασταν από την κατάσταση όπου ο κόσμος πληρώνεται ε, ε, χωρίς λόγο πριν από δύο-τρεις ε, ε, δεκαετίες. Αυτές οι ανισότητες όμως με τη βάση αυτά τα προγράμματά σας δεν θα, δεν θα αγυρωθούν. Γιατί ακόμα και αν δεν λάβουμε υπόψη το κόστος εργασίας και έχουμε αυτό το ανώτατο όριο 100.000 και 60.000, όταν όμως λάβετε υπόψη και το κόστος εργασίας, σίγουρα δεν θα μείνει τίποτα για να μοιραστεί. Η ερώτηση που έχω είναι Μήπως έχει υπάρξει μία οποιαδήποτε δυνατότητα ε, να κερδίσουμε αυτή την, τον αγώνα γιατί ο κόσμος όπως και εγώ που δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα αν δείτε ότι την ανώτατη, το ανώτατο όριο 60 με 100 χιλιάδες οι πυρογνώμος λένε δεν θα μείνει τίποτα για ανακατονομή μήπως είναι μια ψευδής μάχη μια, που δεν έχει κανένα νόημα γιατί ακόμα και αν την κερδίσουμε δεν θα μείνει τίποτα για να ανακατανεμηθεί και τώρα, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Μέγκελ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, uh, uh Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο για να απαντήσουμε σε μερικά σχόλια που έκαναν και οι εμπειρογνώμονες αλλά και τα μέλη της Επιτροπής σας. Καταρχήν και οι τρεις ομιλίες ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και μας ενέπνευσαν και πραγματικά ε, χύνουν φως στο θέμα της κοινής πολιτικής και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής. Συμφωνώ ε, με τον κύριο Χόλονιλ που πολύ εύστοχα και σωστά επισήμανε τις εντάσεις που παρατηρούμε και τις αντιφάσεις μερικές φορές μεταξύ των διαφόρων στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής που θα πρέπει να επηρεάζει το γεωργικό εισόδημα, να λαμβάνει υπόψη το γεωργικό εισόδημα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σωστά στοχοθετημένη προς το γεωργικό εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Θα πρέπει κάπου να είναι απλή, αλλά και δίκαιη ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο να συνδυάσουμε αυτούς τους στόχους. Επίσης δύσκολο είναι να βρούμε την ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των ζητουμένων, αλλά η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή ακριβώ τη δύσκολη ισορροπία προσπαθεί να εξεύρει. Και συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε, διαφορετική, ε, σε διαφορετικό συμπέρασμα για το ποια είναι η σωστή ισορροπία και ίσως θα πρέπει επ' ευκαιρία τη συζήτηση για τη μεταρρυθμίση να σκεφτούμε αυτές τις εντάσεις μεταξύ των διαφορών στόχων να δούμε τα άκρα εντός των οποίων κινούμαστε και να διαρωτηθούμε ποια είναι η σωστή ισορροπία. Αντί να τα βλέπουμε όλα α, και να τα χωρίζουμε σε άσπρο και μαύρο και μερικοί να προτιμούν το άσπρο και μερικοί να, το, να προτιμούν το μαύρο, δεν θα πρέπει να είναι τέτοια η προσέγγιση μας και να μην είναι μεροληπτική η μονομερής. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις και νομίζω ότι αυτό είναι πιο παραγωγικό και επικοδομητικό. Δεν θα επεκταθώ πολύ στα σχόλιά μου. Κύριε Έργιαβετς, είπατε ότι η νέα πολιτική ε, διονύζει τις αδυναμίες του παλιού συστήματος. Δεν συμφωνώ μαζί σας, γιατί τα διαρθρωτικά στοιχεία του προτινόμενου συστήματος είναι ε, αρκετά διαφορετικά από το υπάρχον σύστημα. Είναι ριζικά διαφορετικά. Έχουμε ένα σύστημα σήμερα που οι βασικοί κανόνες ε, αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χωρίς ευελιξία, χωρίς ελαστικότητα και χωρίς τη διακριτική ευχαίρεια που δίνουμε σήμερα με τη νέα πρόταση. Και αυτά εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς ε, περαιτέρω ανάμειξη του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα πρόταση προβλέπει ένα σύστημα όπου σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεσπίζονται λιγότεροι κανόνες και με ορθολογικό διάλογο και ορθολογική συζήτηση με τα κράτη-μέλη και με ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, απειλών και ευκαιριών καταλήγουμε σε ανάλυση των αναγκών και σε στοχευμένα αποτελέσματα με πολύ μεγαλύτερη ελαστικότητα, χωρίς όμως να διαστρεβλώνουμε τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Χρησιμοποιούμε τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ε, στη νέα μας πρόταση και πολύ διαφορετικό μοντέλο. Δεν μπορείτε λοιπόν το, το ισχύον σύστημα να το προβάλλεται στο μέλλον. Γιατί έχει μεγάλες διαφορές. Μιλήσατε ε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στην όλη διαδικασία. Αυτό το προτείνουμε και εμείς. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό τα προγράμματα αυτά να μην χαράζονται σε γραφειοκρατικό επίπεδο, αλλά η κοινωνία των πολιτών, οι δημόσιες αρχές, οι οργανώσεις, ενώσει παραγών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να έχουν και αυτές το λόγο τους στην όλη διαδικασία. Και αυτό το βρίσκεται και στην νομοθετική μας πρόταση. Επίση μιλήσετε για την ανάγκη για τεχνική αρρωγή και γενικώ ε, κάποια βοηθή. Η δυνατότητα τεχνικής αρρωγής προβλέπεται σε επίπεδο 4% από, τον πυλώνα, από το δεύτερο πυλώνα. Είναι διόλου αμεληταίο αυτό το ποσό. Επίσης το ίδιο ισχύει για τη διαδικασία που οδηγεί στην υιοθέτηση των στρατηγικών σχεδίων. Οπότε υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για τα θέματα αυτά. Δεν πιστεύω κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Γιατί θα πρέπει τότε να εξηγήσουμε στους γεωργούς γιατί μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις τους. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να επενδύουμε σε Γραφείοκρατικέ διαδικασίες ή διαδικασίε έγκριση ή προγραμματισμού. Δεν είναι αυτό το σωστό επιχείρημα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία. Ο κύριος Γιώργος Νίλ. άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε για την ισότητα, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει ένα πιο ισότιμο σύστημα. Τι ακριβώς σημαίνει ισότητα στην περίπτωση αυτή. Ο κύριος Φλάναγκαν αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και είπε ότι ίσως στη τελική ανάλυση δεν γίνουν αλλαγές ως προς τους μηχανισμούς στα εργαλεία που προτείνουμε. Αλλά πιστεύω ότι παρά είναι απεσιόδοξο αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σύστημα με ανώτατα όρια, ένα σύστημα κάπινγκ. Έχουμε προαιρετικό σύστημα και πολύ περιορισμένο εφόσον εφαρμοστεί. Και έχουμε τι αναδιανεμητικές πληρωμές που επίση είναι προαιρετικέ για τα κράτη-μέλη. Στο μέλλον θα είναι υποχρεωτικέ, Το ίδιο και τα ανώτατα όρια, οι οροφέ, το κάπινγκ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το κάπινγκ θα χτυπησει 56% 50-60% των εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει να χτυπήσει εκείνου, που για λόγους αθέμητους κατά τη γνώμη του νομοθέτη λαμβάνουν υπερβολικά δαψιλές άμεσες ενισχύσεις. Και σε τελική ανάλυση, και ξαναστέλνω τον μπαλάκι σε εσά, ο νομοθέτης θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Γιατί εμείς ήδη τέσσερις-πέντε φορές ε, ε, προτείναμε σε διαφορετικούς κανονισμούς κάτι τέτοιο και δεν προχώρησε, δεν ευωδόθηκε στην νομοθετική διαδικασία. Ε, άλλοι λένε ότι δεν θέλουν το κάπινγκ, άλλοι θέλουν ότι είναι σημαντικό το κάπινγκ. Είδατε τη διαφορά με την κυρία Γκιλέρα. Θα πρέπει να γίνει διάλογος και κάποια στιγμή να ληφθεί και η πολιτική απόφαση από τους νομοθέτες. Επίσης, η οροφή, το κάπινγκ μπορεί να είναι αποτελεσματικό και εύκολο για διαχείριση, γιατί ο κανονισμό κάνει αυτό που προτείνεται, κύριε Χόγκερνελ. Γιατί προτείνει ε, τους, με, τους τους ε, μηχανισμούς υπολογισμού για τους μισθούς. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετική η μισθή, αλλά αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ένα στάνταρ μοντέλο ε, που το χρησιμοποιούν που συνδυάζει την ε, εργατική δύναμη με τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής δραστηριότητας. Συνδεδεμένες ενισχύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οι συνδεδεμένες ενισχύσεις να περιορίζονται στο 10%, σε λιγότερο ποσοστό από ό,τι σήμερα δηλαδή. Και νομίζω ότι, όπως είπατε, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις παρά είναι γενικές, οπότε όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό τους, τόσο λιγότερο γενικές γίνονται και θα είναι και πιο εύχριστες στη διαχείριση. Οπότε συμφωνώ μαζί σε επίσης έχουμε κάποια όρια σε ό,τι αφορά την παραγωγή και ήδη είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα σήμερα. Νέοι αγρότες. Είναι αγρότες. Αυτό που προτείναμε, κυρίως για την στοχοθέτηση, αυτό που βλέπουμε από τα στοιχεία είναι ότι η... αλλάζει ε, η κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών ό,τι αφορά τη μέση ηλικία των γεωργών. Σε κάποιε χώρε η κατάσταση είναι τραγική. Οι περισσότεροι γεωργοί είναι ηλικιωμένοι. Ενώ σε άλλε χώρε υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ νέων και ε, πιο ηλικιωμένων γεωργών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε και στα κράτη-μέλη την ευκαιρία ε, να προσαρμόσουν τα μέτρα τους για τους νέους γεωργούς ανάλογα με την κατάστασή τους. Οπότε σε ένα κράτος που κατάσταση δεν είναι ανησυχητική να μην αφιερώνονται τεράστια κονδύλια όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Για τη διαχείριση κινδύνου. Σας επισημαίνω τη στρατηγική προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Αυτό που θα θέλαμε στις προτάσεις είναι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν κάτι, ενώ σήμερα τίποτα δεν ε, επιβάλλεται Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς ε, λογικά ανάλογα με τις ανάγκες και την, ανάλυση των αναγκών τους και μετά να κάνουν ό,τι μπορούν στο γενικό στρατηγικό πλαίσιο που θα δημιουργήσουν. Σε κάποιες περιφέρειες και κράτη-μέλη, ήδη με βάση τις, τις κρατικές ενισχύσεις, υπάρχουν κάποια ε, εργαλεία διαχείρισης κινδύνων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα εντάξουμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο που εμπίπτει στο στρατηγικό σχέδιο. Ο πρώην συνάδελφος και φίλος Τόμας Γκαρσία Καράτε αναφέρθηκε σε πολλά στοιχεία του κανονισμού Omnibus. Όντως, εκεί πολλά θέματα από αυτά που είπατε περιλήφθηκαν. Είπατε ότι ο έλεγχος δεν θα πρέπει να είναι αναδρομικός. Μα εξορισμού είναι αναδρομικός ο έλεγχος. Είδατε τι συνέβη στο παρελθόν. Αναλύει μια κατάσταση του παρελθόντος και αξιολογεί την κατάσταση αυτή με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, είτε της ανάκτησης ε, κονδυλίων, είτε της διόρθωσης των ε, Τη χρηματοδότηση επίση έχουν αναδρομική ισχύ, γιατί ο έλεγχος εκφύσεω εξετάζει κάτι που συνέβη στο παρελθόν, αυτό δεν αλλάζει. Διαφάνεια των τιμών. Ναι, παραλάβω αυτό που σας είπα και την περασμένη φορά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια στις τιμές. Θέλουμε να βελτιώσουμε του μηχανισμού που ήδη ισχύουν στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού ή στα πλαίσια των αθέμητων εμπορικών πρακτικών τώρα, ώστε οι γεωργοί να γνωρίζουν καλύτερα για την κατάσταση των τιμών στην αγορά. Έτσι θα αντιληφθούν καλύτερα πού απορροφούνται τα μερίδια της προστιθέμενης αξίας στην διατροφική αλυσίδα. Θα εκπονήσουμε και μία μελέτη αντικτύπου. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε τη διαδικασία στα πλαίσια των κατεξοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Για την κρίση, Τόμας, είπες ότι χρειαζόμαστε κριτήρια που θα ενεργοποιούν ε, τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια γενική ρήτρα στον κανονισμό για την ΚΟΑ. Άρθρα 2.19, 2.21 και 2.20 για φυτογενομικές κρίσεις και επιζωτίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν εν ανάγκη. Και προτιμούμε αυτή τη γενική ρήτρα, γιατί ο σαφής προσδιορισμός των κριτήριων μπορεί να αποτελέσει ανοιχτή πρόκληση για την πυροδότηση μέτρων κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να εξετάζουμε τη γενική κατάσταση της αγοράς, την συνολική κατάσταση σε ό,τι αφορά το γεωρικό εισόδημα, τη διαπραγματευτική θέση στην διατροφική αλυσίδα και κάποια στιγμή να ε, εξακριβώνουμε κατά πόσο όντως υπάρχει ανάγκη για την ανάληψη δράσης. Γιατί η ανάληψη δράση δεν είναι μόνο θέμα καλής βούλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι και θέμα προϋπολογισμού. Και όπως είδαμε και στο παρελθόν, είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια για να έχει νόημα με τέτοια δράση. Και αυτό σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει το μέλλον. Σε ό,τι αφορά αυτά τα ραδίκια αντίβ, ίσως το πρέπει να το συζητήσουμε διμερώς για το κατά πόσο μια οργάνωση παραγωγού από μόνη της είναι ξεχωριστή οικονομική οντότητα με βάση το δίκαιο ανταγωνισμού. Ίσως εκεί δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Πάντως συμφωνώ με το άρθρο 152, όπω προκύπτει από τον κανονισμό Omnibus, ότι με βάση αυτό το άρθρο είναι δυνατόν πια να εξαιρούνται ζωτικέ δραστηριότητε οργανώσεων παραγωγών από τις ε, διατάξεις του ανταγωνισμού. Αρκεί να έχουν κάποια οικονομικά πλεονεκτήματα. Δεν μιλούμε μόνο για διαπραγμάτευση, αλλά για να ε, ολοκληρώσουν τις οικονομικές δραστηριότητες των μελών τους. Για τη διαχείριση των κρίσεων αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια. Οπότε υπάρχει δυνατότητα ε, να έχουμε επιχειρησιακά προγράμματα και σε άλλους τομείς πλην των απορροκυπευτικών. Κύριε Καλινόφσκι, μιλήσατε στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει για το κατά πόσο θα λαμβάνουν οι γεωργοί άμεση ενίσχυση όχι. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό που λέει η πρόταση είναι ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα παραμείνουν θεμελιώδη στοιχείο ε, στήριξη του γεωργικού εισοδήματο και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προγραμματίζουν ή να σχεδιάζουν τις άμεσες ενισχύσεις που θα χορηγούν στα πλαίσια των στρατηγικών του σχεδίων. Και αυτά τα στρατηγικά σχέδια εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι ουρανοκατέβατα, όχι αυθαίρετα, αλλά με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια που περιλαμβάνει η πρόταση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να αποφασίσει από μόνη της, από το κεφαλιού της αν θα λαμβάνει ο Γιώργος άμεσες ενισχύσει. Οι άμεσες ενισχύσει θα εξακολουθούν να είναι η ραχοκοκαλιά της κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης αναφέρθηκαν σε κάποια σχόλια ε, τα θέματα της σύγκλησης και ότι υπάρχει μια φαιά ε, και κάποιες ε, παρεξηγήσεις για το νόημα της σύγκλησης. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ώστε οι στραματικές ενισχύσεις που δίνονται στα κράτη-μέλη, καλό θα είναι να συγκλίνουν όσο γίνεται, ώστε όλοι όσοι έχουν στραματικές ενισχύσεις κάτω των 200 ευρώ ανά εκτάριο, θα αυξηθούν, ώστε να υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ των ενισχύσεων. Και αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα μεταξύ παλιών και νέων χωρών μελών και σε παλιέ χώρε μέλη υπάρχουν διαφορές στο ύψο των στρεματικών ενισχύσεων. Μερικές φορές είναι σε ένα τμήμα μόνο του κοινοτικού μεσόρου, στο 90% του κοινοτικού μεσόρου και θα υποφεληθούν από αυτή την σύγκληση. Υπάρχει επίση το 75% αλλά αυτό δεν ισχύει για τα νέα κράτη-μέλη. Για τα νέα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ένα υποσύστημα που είναι κατά με το ίδιο ποσοστό ανά εκτάριο. Οπότε τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά ακόμη ε, δικαιώματα εφαρμόζοντας τις ιστορικές αναφορές για το σύστημα θα πρέπει τις αξίες των ε, διαφορετικών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να τις φέρουν πιο κοντά. Θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση στο ύψος των ενισχύσεων. Δεν θυμάμαι απ' έξω το άρθρο, θα σας το πω αργότερα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη αυτά να μεριμνήσουν ώστε το ελάχιστο επίπεδο της αξίας του δικαιώματος να φτάσει στο 75% του εθνικού μεσόρου. Αυτό είναι εσωτερική σύγκληση και δεν έχει σχέση με τα νέα κράτη-μέλη, γιατί εκεί ισχύει το καταποκοπή ποσό. Ε, τα κράτη-μέλη όμως, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία που εφαρμόζουν το, τα ιστορικά κριτήρια, θα ε, πρέπει να επηρεάζονται από το νέο σύστημα. είπατε, ε, αναφέρατε ότι θα υπάρχουν τα ίδια μέσα στους δύο πυλώνες. Αυτό που βρίσκεται στην πρόταση είναι ότι θα υπάρχουν ε, γεωργοπεριβαλλοντικά συστήματα στις διάφορες ε, μεταβλητές τους, όπως ήδη συνυπάρχουν σήμερα. Τα μέτρα αυτά θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, να είναι εφαρμοστέα θα, ε, τα ακολουθούν τα κάτι μελη που θα ακολουθούν και τα κριτήρια του στον κανονισμό. Αυτό όμως που σημαίνει αυτό για τον πρώτο πυλώνα είναι ότι τα κάτι μελη θα μπορούσαν 100% να χρηματοδοτήσουν από τον Ευρωπαϊκό Νόμο και να αναπτύξουν πολύ στοχοθετημένα, ακόμα πιο στοχοθετημένα συστήματα από ότι ε, στο γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα για ανάλογα με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα που έχουν στη δικιά τους επικράτεια. Δεν, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν 5, 10, 15% του προπολογισμού τους γι' αυτό, να πάρουν όμως θα μπορούν το μερίδιο που θεωρούν ότι είναι ε, κατάλληλο. Και όπως είπε και κάποιος από τους εμπειρογνώμονες, τότε τα κρατημέλη θα μπορούσαν όχι μόνο για παράδειγμα να πληρώνουν ε, τα εισόδημα και τα επιπλέον κόστη, αλλά να συμπεριλαμβάνουν και ένα στοιχείο κινήτρου που από ό,τι κατάλαβα είναι ένα ε, ευρέως δεδομένο αίτημα εδώ σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και εκτός ε, στην ε, κοινότητα των Γεωργών. Είναι ένας τρόπος λοιπόν για να δοθεί στα κράτη-μέλη ένα επιπλέον μέσο για πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνεται στο στρατηγικό του σχεδιασμό και έτσι θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει επιπλέον διοικητικός φόρτος. Τέλος, ε, Πάλι εσείς κύριε Καλινόφσκι νομίζω είπα, αναφέρατε το άρθρο 4 και το 16 αυτή η περίφημη ρήτρα για το γνήσιο αγρότη που έχει πολύ επικριθεί, τον πραγματικό αγρότη, και να αναφέρατε μια περίπτωση στη χώρα σας όπου οι αγρότες μπορεί να μην μπορούν να ε, διεκδικήσουν ε, στήριξη των τιμών που μάλλον καταβάλλεται από το εθνικά κονδύλια, αυτό έχω καταλάβει, διότι δεν έχουν ε, τις εκτάσεις υπό τον έλεγχό τους. Εγώ θα έλεγα ότι για αυτή την περίπτωση θα πρέπει ίσως να κάτσουμε μαζί και να εξηγήσετε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα για να δούμε αν πρόκειται για πραγματικό πρόβλημα για την επιτόπου εφαρμογή των μέτρων των κοινοτικών. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να έχουμε και σε επαφή με τις πολωνικές αρχές για να δούμε αν κάτι πάει στραβά ή αν είναι απλά μια συνέπεια που παίζει ρόλο στο πλαίσιο της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων όπου η Κομισιόν δεν είναι πραγματικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή. Αυτά λοιπόν έχω να πω, και υπήρχαν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, αλλά νομίζω πως ήδη έχω αναλύσει αρκετά το θέμα. Ναι, σχεδόν πέρασε στο 21ο λεπτό της παρέμβασής ναι. σας. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Αν και δεν λύσατε το πρόβλημα του κύριου Καλινόφσκι. Αυτά είναι εσωτερικά θέματα, είναι ζητήματα της Πολωνίας. Ο κύριος Καλινόφσκι. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι όντως περίπλοκο το, προ, το θέμα. Ούτε σχεδόν και εσείς δεν καταλάβατε το πρόβλημα που ε, επισήμανα και ο κύριος Διευθυντής ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εγκρίνει τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα ήθελα να να ασχολείται με τους πραγματικούς ενεργούς γεωργούς γιατί αναφέρονται οι ορισμοί που γίνονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμοι αυτοί οι ορισμοί γιατί στην Πολωνία δεν λαμβάνει μόνο ο πραγματικός γεωργός άμεσης ενισχύσης πάνω από τις μισές άμεσης ενισχύσεις στην Πολωνία δίνονται σε ε, δικαιούχους που δεν είναι γεωργοί ξέρετε και εσείς από μόνος σας ε, ε, το, το πρόβλημα ναι, ναι, αλλά δεν το γνωρίζουν όλοι αυτό. Παρακαλώ, οι πυρογνώμονές από 10 λεπτά ο καθένας. 10 λεπτά το πολύ ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σλοβενικά για αλλαγή. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, με κάποιους ορισμούς βασικούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μία φάση στρατηγικού σχεδιασμού για την κοινή γεωργική πολιτική της. Ε, αυτό είναι κρίσιμο, γιατί στο παρελθόν κάναμε διάφορα πράγματα χωρίς να γνωρίζουμε το μέλλον. Τι είναι ο στατηγικός σχεδιασμός, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας με βάση επιστημονικά δεδομένα, επιστημονική ανάλυση και όχι με βάση ε, ορισμένες ομάδες συμφερόντων που ισχυρίζονται διάφορα πράγματα ότι ισχύουν γιατί έτσι αντιμετωπίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και έτσι είμαστε σε θέση να βρούμε και τους σωστούς στόχους. Η καλή πολιτική βασίζεται σε μετρήσιμους στόχους, ποσοτικοποιημένους. Και εκεί θα πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά ε, μέσα στο παρόν, στο ισχύο νομοθετικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο τα κατάλληλα μέτρα για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δύο είναι λοιπόν εδώ τα προαπαιτούμενα για να είναι σωστός και επιτυχής ο σχεδιασμός. Πρώτον, ποιοτικός έλεγχος, σαφές αυτό, και ε, δεύτερον να αποφύγουμε όσο γίνεται να βάζουμε ε, διάφορα ιδεολογικά εμπόδια, ιστορικές καταβολές, χειραγώγηση λόγω συμφερόντων κλπ. Μόνο έτσι θα υπάρξει μεταρρύθμιση και με στρατηγικό σχεδιασμό. Χωρίς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να ε, συμμετέχουν εκπρόσωποι ε, των γεωργών, εκπρόσωποι οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και λοιπόν που μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις ε, ως προς τον επιθυμητό στόχο και αποτέλεσμα. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας λοιπόν. Και με βάση αυτές τις ε, αρχές και τις προτάσεις προσπαθώ να απαντήσω στα όσα ρωτήσατε. Πρώτη ερώτηση μάλλον πρώτη απάντηση, είναι προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μέγκελε. Για την πλήρη αλλαγή πορείας της κοινή γεωργικής πολιτικής και ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι τεράστια αλλαγή και το θεωρούμε προβληματικό το γεγονός ότι μεταφέρεται από το δεύτερο πυλώνα πάρα πολλά θετικά αλλά και αρνητικά, που είναι τα γενή σφάλματα της σημερινής πολιτικής. Η πολιτική αυτή είναι πάρα πολύ ήπια, πάρα πολύ soft. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και αντικειμενικοί στόχοι όσοι θα όφυλαν όταν σχεδιάστηκε. Άρα αυτό συνδέεται και με την ίδια την ποιότητα των διοικητικών ε, διαδικασιών. Και ποιο είναι εδώ το βασικό πρόβλημα με την κοινή μας ε, πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη και το στρατηγικό σχεδιασμό. Ότι οι ανάγκες αυτές δεν είναι όσο σημαντικές θεωρούμε εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει ο προπολογισμός η αναδιανομή των κονδυλίων κτλ. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει βασιστεί σε μία ανάλυση ε, ήπια. Αυτό είναι ένα πρωτόγωνο εργαλείο για μένα. Είναι αβέβαιο, είναι ανασφαλές, είναι αναξιόπιστο και δεν μας οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλες μας λοιπόν οι προτάσεις αφορούν αυτό, ότι θα πρέπει οι στόχοι να είναι μετρήσιμη Και εκεί χρειάζεται διόρθωση όλων των στρεβλών του παρελθόντος. Εκεί συνοψίζεται για μένα η σημερινή συζήτηση. Πρώτον, όπου υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πρέπει αυτή να συνδέει ε, τους στόχους και τα μέσα και τα μέτρα με πραγματικές αναφορές στην κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή, τι εννοώ. Κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, ε, Αυτά θα πρέπει να τα συνδέουμε. Προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των υδάτων, προστασία των εδαφών. Όπου υπάρχει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για όλα αυτά, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχουν βρεθεί οι άμεση σύνδεσμοι και οι άμεση σχέση. Εάν ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι οι στόχοι μας και πού θέλουμε να πάμε με την εκάστοτε πολιτική, θα πρέπει να συνδέονται αυτά και να καταλήγουμε σε μεμονωμένα επιχειρησιακά σχέδια. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με το εισόδημα των γεωργών. Αυτό είναι κομβικό στην κοινή γεωργική πολιτική και θα παραμείνει. Και δεν είμαι σίγουρος ότι με τη νέα πρόταση αλλάζει αυτό. Οι νέε προτάσεις δεν μιλούν για επίπεδα εισοδήματος, ούτε για το ε, ποιο είναι οι δικαιούχοι και ποιοι είναι οι ομάδες στόχοι. Αυτό μπορεί να οριστεί με κάποιο τρόπο στις Βρυξέλλες και μετά να μπουν τα κράτη-μέλη και να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά με άλλο τρόπο. Τα μέτρα και τα ε, κονδύλια που δεν έχουν κατανεμηθεί στο παρελθόν με δίκαιο τρόπο. και αυτός που θα μπορεί να δικαιολογήσει τα έξοδά του μπορεί να βραβευτεί και με το βραβείο Νόμπελ. Λοιπόν, το πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι στους αγρότες δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν γίνεται χωρίς υποστήριξη. Και γιατί κάποιοι θα πρέπει να υποστηρίζονται και κάποιοι όχι. Και γιατί να τα αποφασίσουν οι Βρυξέλλες. Δεν μπορούν να τα αποφασίσουν αυτά οι Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να λυθεί. Ε, ε, και τώρα, για το στρατηγικό σχεδιασμό, ε, και αυτός έχει να κάνει με την νομιμοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αν κανένας δεν την πιστεύει την κοινή γεωργική πολιτική στην πράξη, γιατί θέλουν όλοι να διατηρηθεί και την υπερασπίζονται. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν, ούτε πολιτικό, ούτε αγρότη, ούτε κανένα που είναι 100% ικανοποιημένο. Αλλά κανεί δεν θέλει και να καταργηθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Και αν είναι στα χέρια των κρατών μελών, αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία ενδεχομένω. Να βγάλουμε κάτι από την πολιτική αυτή και να αποφύγουμε, θα είχαμε αποφύγει το Brexit και όλα αυτά. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να ε, χρησιμοποιήσουμε σωστά το στρατηγικό σχεδιασμό. Κάποιος είπε ότι θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε κάθε ε, πιθανή και απίθανη ε, ένωση και οργάνωση παραγωγών. Ε, να γίνεται καλός στρατηγικό σχεδιασμός όχι από κάποιες κεντρικές διοικησει στα κράτη-μέλη αλλά με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων των γεωργών, των περιβαλλοντολόγων, των ε, ε, οικολόγων, των ενδιαφερομένων. Ενδιαφέρον είναι αυτό και δημιουργικό αλλά δεν είναι η διοικητική πρακτική. Και τι... Θυμήθηκα τώρα κάτι σε σχέση με το κράτος μέλος το οποίο προεδρεύει αυτό το καιρό στο Συμβούλιο. Και κατάλαβα γιατί είναι τόσο πρόθυμη η Αυστρία να εξετάσει το θέμα. Όταν εμείς στη Σλοβενία ε, υιοθετήσαμε αυτή την πολιτική μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι ψάχναμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Και είναι ένα καλό παράδειγμα. Και θα μπορούσαν όλα τα κράτη-μέλη και ε, όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να συνεργαστούν και να προσπαθήσουν να λύσουν αυτό το θέμα και να ε, διευκρινιστεί πού πηγαίνουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, αυτός ο χορός των δισεκατομμυρίων. Και για να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που μου έγιναν προηγουμένως, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να αποφύγουμε να υπάρχει ένας εργαζόμενος, ένα γραφείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να χειρίζεται το θέμα μόνος του. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ ευρύ το πεδίο και θα πρέπει η ποιότητα των ε, διαδικασιών λήψεων αποφάσεων να βελτιωθεί με τη σωστή εμπειρογνωμοσύνη έτσι ώστε όλα αυτά να έχουν επιτυχή έκβαση. στο στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει να συμμετέχουν οι πάντες. Και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν το ρόλο τους. Αλλά είναι σαφές ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσουν, γιατί παρακολουθεί τη διαδικασία ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ποιότητά της. Και εκεί μπορεί να ακούσει ενεξάρτητους φορείς, think tank από τα κράτη-μέλη. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε ή όσο θα μπορούσαμε. Ευχαριστώ. Είπα 10 λεπτά το πολύ ο καθένα. Okay, I would, I would like to address a, few Θα ήθελα να... απαντήσω σε κάποια σημεία και στα θέματα τα οποία διευκρίνησε η Επιτροπή ο συνάδελφος εγώ δεν θα μπω. Καταρχάς λοιπόν η παρατήρηση κυρία Ροντρίγκε για το κατά πόσο η πολιτική θα πρέπει να κατευθυνθεί περισσότερο προς την κατεύθυνση των τιμών. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο και δεν ήταν πρόθεσή μου να του πω κάτι τέτοιο άμεσα. Πάντως, αν δείτε ότι έχουμε περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά πολιτική, θα θέλαμε να έχουμε και κατευθύνσεις από την αγορά. Από την άλλη πλευρά θα έλεγα πως αυτή η αρχή είναι κάτι που ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί έτσι η Γεωργία θα μπορούσε να συμβάλλει και στο θέμα της ε, γενικότερης κατάστασης της, ε, των τροφίμων παγκοσμίω. Τώρα, αν έχουμε πολύ ψηλέ ε, απαιτήσει όμως αλλού, που δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν, ας πούμε, από την αγορά, τότε θα έπρεπε να δούμε ένα περισσότερο κάποια μεγαλύτερη απέτηση ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί ένας γεωργός που έχει μεγαλύτερες απαιτήσει να παίξει και ρόλο στο περιβάλλον της αγοράς. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ήδη είπε ότι η πρόταση επιτρέπει να συμπεριληφθεί μια ρυθμιστική, ένας ρυθμιστικός υπολογισμός για τα εισοδήματα, ας πούμε. Ναι, αυτό το βλέπω και εγώ. Αλλά εγώ έλεγα να προχωρήσουμε και κάπως περισσότερο, να υπάρχει και ένας ρυθμιστικός υπολογισμός ε, σε σχέση με την εργασία αναεκμετάλλευση. ερώτηση τώρα του κυρίου Φλάναγκαν για την ανακατανομή. Είπατε ότι το κάπινγκ ε, ακόμα και αν ε, αλλάξει το επίπεδο ε, δεν θα αποφέρει τα χρήματα ώστε να μπορέσει να γίνει ανακατανομή. Νομίζω πως γι' αυτό συμφωνώ, αλλά αυτό δεν αποκλείει το κράτος μέλος από την ανακατανομή πληρωμών ή χρημάτων. Okay. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. In itself, they say the, the uh, unequal distribution of the, of the, of the payment, that's... Uh, Αυτό το ίδιο σημαίνει μια άνηση κατανομή των πληρωμών. Αυτό το, έρχεται από το παρελθόν, γιατί έχουμε στήριξη των τιμών, που ευνοεί τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και μετά έχουμε τις πληρωμές ανακτάριο που η ίδια βάση καταρχήν και οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και πέρα ακόμα πιο στοχοθετημένη του προγράμματος. Υπήρξε και η παρατήρηση για την ισότητα. Για την ισότητα που τη χρησιμοποίησα χωρίς να καταστήσω απόλυτα σαφές τι εννοούσα. Συμφωνώ γι' αυτό. Όταν μιλάμε για ανισότητα, λέμε ναι, 80% των πληρωμών γεωργίας πάνε στο 20% των γεωργών. Αυτή είναι μια σαφής ανισότητα. Όμως όταν ρωτήσει κανείς πώς θα τα κάνουμε καλύτερα, τότε χρειάζονται καλά κριτήρια. Γιατί ε, μια μεγάλη εκμετάλλευση απασχολεί πολλούς εργαζόμενους. Άρα αιτιολογείται. Και υπάρχουν και αποδείξεις από διάφορες μελέτες και από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται η στήριξη για, ορισμέ, για κάποια εκμετάλλευση, ενώ υπάρχουν άλλες που μπορεί να χρεια... το... τη χρειάζονται στήριξη περισσότερο από αυτή που παίρνουν. Πρέπει να βρούμε κάποια τυπικά κριτήρια αριθμιστικά. Έκανα μια τέτοια πρόταση να κατευθυνθούμε προς τα εκεί, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη και αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, να μην τα βλέπουμε άσπρα μαύρα τα πράγματα. Και η δική μου πρόθεση αυτό ήταν να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει τελείως να ανατρέψουμε το σύστημα. Για την συνδεδεμένη στήριξη εισοδημάτων συμφωνώ εάν μειωθεί το σύνολο του ποσού που μπορεί να χορηγηθεί μπορεί να έχουμε αυτό το, τον αντίκτυπο. Δεν είναι ίσως τόσο δύσκολο. Έχω εδώ όμως κάποιες ε, ανησυχίες τις οποίες έχω εκφράσει. Διαχείριση κινδύνου, να το δούμε αυτό σε ευρύτερο πλαίσιο. Νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό και η πρόταση αυτό το προβλέπει. Και θα ήθελα να προτείνω, ναι, να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε το ίδιο επίπεδο. Για παράδειγμα, αν δούμε στη Γερμανία πώς οργανώνεται η διαχείριση κινδύνου, χρησιμοποιείται ο ιδιωτικός τομέας, ενώ σε άλλες χώρες ίσως η ισορροπία να κρατιέται με άλλο τρόπο. Υπάρχει μια ιστορία δηλαδή εφιστάμενων συστημάτων. Δηλαδή να μην τα ξαναστήσουμε όλα από την αρχή τα συστήματα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συστήματα που υπάρχουν. Τώρα για το οίκο σχήμα. Αυτό που σκέφτηκα ότι θέλουμε να έχουμε βάση περισσότερο τα αποτελέσματα, την απόδοση. Κατά τη δική μου γνώμη, είναι δυνατόν να περιλάβουμε και διάφορα συστήματα. Το σύστημα ε, πόντων θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει μεγαλύτερη συμμετοχή. Εγώ θεωρώ πως είναι κάπως ευρύτερο. Δηλαδή, λέει η Κομισιόν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει κάποια χώρα. Εγώ πιστεύω πως θα μπορούσε να είναι γενικότερο σύστημα για να την επίλυση γενικότερων προβλημάτων. Ας πούμε, για τις συνθήκες και για τις περιβαλλοντικές πρακτικές. Ε, είπατε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας χώρος ε, ε, buffer 10 μέτρων ή 20 μέτρων. Αυτό μπορείς να κάνεις στο 20 σκιμ, να βάλεις τα επιπλέον 10 μέτρα εκεί. Κάποιοι γεωργοί το κάνουν αυτό, κάποιοι όχι θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει. Επίση, μέσα σε αυτό το οικοσκήμο, όταν αμείβει κάποιου ε, γεωργού επειδή κάνουν κάποια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, μπορεί αυτό να τους δώσει κίνητρο και επιχειρηματικό. Ναι, τα περιβαλλοντικά προγράμματα μπορούν να το κάνουν, τα έχουμε στο δεύτερο πυλώνα. Ναι, μπορούν, αλλά υπάρχει ένα περιορισμό στην πληρωμή και τονίστηκε αυτό. Ενώ στο οικοσκήμ μπορείς να έχεις ψηλότερη αποζημίωση με κάποιο κέρδος και σημαίνει πως είναι πιο ελκυστικό για να συμμετέχει κανείς. Και το έχω αυτό κάπως στο μυαλό μου. Ότι δηλαδή μέσα των 20 θα είχαμε ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα με μεγαλύτερη συμμετοχή από τους γεωργούς, ενώ στο δεύτερο πυλώνα έχουμε τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα για πιο ε, βαριά μέτρα που δημιουργούν μεγαλύτερη προσπάθεια για τον γεωργό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, το γεωργικό εισόδημα, εγώ πρότεινα αφενός να αναθεωρηθούν οι ενδεικτικές τιμέ για να προσαρμοστούν στις πραγματικές συνθήκες αγοράς και να επιτρέψουμε την ιδιωτική διαχείριση ως προληπτική διαχείριση. Δεν κρίνω σκόπιμο να επιστρέψουμε στο προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στην αγορά και στις μηνιαίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία επιδότηση έχει μετατραπεί σε μεγάλο εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων. Στην Ισπανία το 50% της τελικής γεωργικής παραγωγής εξάγεται εκτός της Ισπανίας. Ένα τμήμα πηγαίνει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα άλλο σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα βγει κερδισμένη από τον προσανατολισμό στην αγορά, αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους μηχανισμούς ώστε να επιτρέπεται πιο εύκολη παρέμβαση στην αγορά. Επίσης, κάποιοι μηχανισμοί διαχείρισης ε, της προσφόρας και αν στους ε, παρόντες κανόνες ε, του Διεθνού εμπορίου υπάρχουν οι μηχανισμοί της προσφοράς, αν περιορίσουμε την ευρωπαϊκή προσφορά, αφήνοντας περισσότερο περιθώριο στις εισαγωγές. Ίσως έτσι αμφισβητήσουμε τις διεθνείς συμφωνίες. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει αποφεληθεί ιδιαίτερα από την απελευθέρωση των γεωργικών αγορών παρά κάποια προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένες ζώνες. Θα συνεχίσω λοιπόν στα αγγλικά τώρα για τις υπόλοιπες απαντήσεις. Στην πρότασή μου να γίνει συγχώνευση του 10% της ενδεδεμένης ε, ενίσχυσης με το 3% της ε, άλλης ενίσχυση, ώστε να φτάσουμε ίσως και σε 20% για τέτοιου είδους ενισχύσεις με βάση την ε, εμπειρία για τα προκυπευτικά το 90% των ενισχύσεων για τους οργανώσεις παραγωγών είναι από το πράσινο κουτί και από Οπότε στηρίζουμε και τις οργανώσεις παραγωγών και ευθυγραμμιζόμαστε με τους κανόνες του ΠΟΕ και στηρίζουμε τα ποροκυπευτικά και τους οργανώσεις παραγωγών. Και καλύτερα να έχουμε συνδεμένες ενισχύσεις ε, που προσανατολίζονται προς το πράσινο κουτί παρά να είναι εκτός. Επίσης, εμείς και τότε δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρώτη κρίση του γάλακτος δώσαμε 200-300 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ για τους γαλακτοπαραγωγούς με αύξηση της άμεσης ενισχύσης χωρίς να επηρεάσουμε την αγορά. Και σίγουρα ο καθηγητής Άλαν το τόνισε αυτό. Επίσης, είναι σαφές για μένα και για το δικαστήριο ότι μια εμπορική οργάνωση παραγωγού δεν είναι καρτέλ, είναι επιχείρηση. Και αυτή ήταν μια συζήτηση που είχαμε με την ε, Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ που ήταν ήμουν στην άλλη πλευρά. Ε, μια εμπορική ε, οργάνωση παραγωγών είναι επιχείρηση και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αν κανείς πιστεύει ότι η οργάνωση παραγωγών είναι καρτέλ, είναι μια δεστραμμένη σκέψη και ο αρνητικός αντίκτυπος μιας τέτοιας αντίληψης ε, πλήττει τη γεωρική κοινότητα. Αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό το σημείο τώρα για τον έλεγχο. Ε, φυσικά ο, ο έλεγχος είναι αναδρομικός, αλλά εγώ είμαι κατά της ε, ε, αναδρομικής ερμηνείας των κανόνων. Έγινε το 2006 μεταρρύθμιση του τομέα των απορροκυβευτικών. Και τότε επιτρέψαμε στις οργανώσεις παραγωγών να αναθέσουν εξωτερικά κάποιες δραστηριότητες. Ήταν σαφές τότε και ως εταιρεία μία οργάνωση παραγών μπορεί να κάνει μια οργανωση παραγωγών μπορει να εξωτερήκευση και να αναθέσει εξωτερικά το σκόπιμο και εσωτερικά τα υπόλοιπα. Αυτό είναι δικαίωμα κάθε επιχείρησης. Ε, βέβαια, η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του ελεγκτή ήταν τελείως διαφορετική. Και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα με τα κράτη-μέλη. Τι συνέβη τότε, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ευελιξία στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη και οι διοικήσεις τους σκέφτηκαν. Τι πρόβλημα θα βρουν οι ελεγκτές σε μία πενταετία. Ως εκ τούτου θα αρχίσουν από τώρα να κάνουν ακόμα πιο περίπλοκες νομοθετικές διατάξεις για να αποτρέψουν αυτό που ενδεχομένω θα έβρισκε πέντε χρόνια μετά ο ελεγκτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό πραγματικά περιπλέκει τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να διαβεβαιώσουμε τις εθνικές ενισχύσεις ότι αν σήμερα καταλαβαίνουν την εξωτερήκευση ω διακριτική ευχαίρεια της επιχείρησης να αναθέσει κάποιες δραστηριότητε εκτός αυτής, Έτσι θα το κρίνει μετά από μία πενταετία και ο ελεκτή όταν έρθει. Όταν θα κρίνει τι συνέβη πριν από πέντε χρόνια. Αν πριν από πέντε χρόνια γνώριζα τι ξέρω σήμερα, σίγουρα θα απέφευγα πολλά σφάλματα. Αυτό ακριβώς ζητούμε από τα κράτη-μέλη, να προλάβουν ουσιαστικά. Αυτό που θα έρθει μετά από μία πενταετία κάποιος και θα κρίνει. Και τι θα σκεφτεί ο ελεγκτής. Αυτό όμως περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Όχι αναδρομική ερμηνεία λοιπόν, όχι αναδρομικός έλεγχος, αλλά είμαι κατά της αναδρομικής ερμηνείας της νομοθεσίας. Επίσης, θα έλουμε μια προβλεψιμότητα σε παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν θέλουμε να έχουμε μια διαχείριση κινδύνου που γίνεται μόνο μέσω ιδιωτικής και δημόσιας παρέμβασης, πλήρω ιδιωτική ή μετερική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην αγορά. Μερικοί κίνδυνοι είναι ε, κλασικοί. Αν θέλουμε ε, να έχουμε ένα πρόγραμμα ώστε να επηρεάσουμε την αγορά ή ένα είδος αμοιβαίας ε, ενίσχυσης, θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι κίνδυνοι ασφαλίζονται, ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, από τα μειολοβοήθειας μάλλον. Το είχαμε πει πριν από καμία διετία που είχαμε έρθει στην Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Γιατί έχουμε τον κίνδυνο στη γεωργική εκμετάλλευση, έχουμε το γεωργικό κίνδυνο. Έχουμε του κλασικού ε, κίνδυνου τη αγοράς, αυτούς τους διαχειρίζεται η οργάνωση παραγωγών ή η παραγωγή. Και έχουμε κίνδυνο που ε, υπόκειται σε ασφαλιστικό συμβόλαιο. Υπάρχει όμω και ένα κίνδυνο ε, αγορά που δεν το γνωρίζουμε. Πότε θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρέμβαση. Και αν δεν ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αν δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα παρέμβει στην αγορά, τότε δεν θα έχουμε καμία ιδιωτική ασφάλιση ή ε, ασφάλιση ταμιόλου βοηθείας ή κοινή ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση. Πώς να μπει κανεί ε, στο παιχνίδι αν δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι κινδύνους θα αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το χειρότερο για, ένα, για μια ασφαλιστική επιχείρηση, ένα ταμείο βοηθείας το να, η αβεβαιότητα ως προς τον κίνδυνο. Θα πρέπει να γνωρίζει τι κίνδυνο ασφαλίζει. Και αν θέλουμε κάποιο είδο ασφάλεια στην αγορά, η ασφάλεια στην αγορά, θα πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους. Αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, καλώς. Αλλά να γνωρίζουμε τότε ότι δεν θα έχουμε καμία ιδιωτική ασφάλιση, κανένα πρόγραμμα ιδιωτικής ή ε, δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Για κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη προηγούμενη γνώση του, του κινδύνου που ασφαλίζεται. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και για την οικονομία που μας κάνατε, για την γενναδορία σας μάλλον. Μας θα χαρίσετε και ένα δίλεπτο. Ευχαριστούμε πολύ για τις ομιλίες και τις απαντήσεις που καταδεικνύουν την περιπλοκότητα αυτού του θέματος. Πάντως σίγουρα εμπλουτίσετε τις γνώσεις, τις γνώσεις μας, αλλά ε, εμπλουτίσατε και τις ανησυχίες μας, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και νομίζω ότι μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας αυτής της δημόσιας ακρόασης. Ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ποια, ποιο είναι το μέγεθος των προκλήσεων σε ό,τι αφορά τη νέα κοινή ορική πολιτική μετά το 2020. Θα πρέπει όμως να ανταπεξέλθουμε και να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Λίγο χρόνος μας έχει μείνει, εξού και ο εντατικός ρυθμός των εργασιών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, τους εμπειρογνώμους, τα μέλη της Επιτροπής και τους ευρωβουλευτές που έλαβα μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, Περνάμε στα διάφορα. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, να κηρύξουμε το πέρας της συνεδρίασης. Έχουμε και συνεδρίαση στο Στρασβούργο 22 Οκτωβρίου. 22 έτσι δεν είναι. Στις 7. Ημέρα Δευτέρα, 7 για 2,5 ώρες ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Άγκρη. Αυτά. Λύεται η συνεδρίαση.